Then with Δεύτερο λοιπόν, δεύτερη συνεδρίαση σήμερα. Κάποιες σύντομες ανακοινώσεις. Να επιστήσω την προσοχή σας στην εκστρατεία του συνδικάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο που λέγεται "Dying to Work, πεθαίνω να δουλέψω σχέση επαγγελματικής δραστηριότητας με τις ασθένειες. Δύο εκπρόσωποι των Βετανικών Συνδικάτων επισκέπτονται σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο ε, with posters and they hope that ε, ε, Employment Committee will θα μπορέσουμε ίσως αν θέλετε να φωτογραφηθούμε σαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Απασχόληση με το πόστερ της εκδήλωσης αυτής, της εκστρατείας αυτής. και να δώσουμε και τη μάχη για να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι διαθέσιμα τα πόστερ για φωτογραφίες ανάμεσα στις 3 και τις 5. Θα ξεκινήσουμε τώρα τις ψηφοφορίες, οπότε όσοι θέλουν να φωτογραφθούν μπορούν να το κάνουν μετά. Έχετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Έχετε επίσης και τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική C αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. B αγγλικό ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F αγγλική ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 17. Πέρα στις ψηφοφορίες. 22 υπέρ, 27 κατά, καταπίπτει. 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 19, ψηφίζεται. Δεκτή. 27 υπέρ, 24 κατά. Ή μπι αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. CA υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ή e υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. HA υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα. 28 υπέρ. Α, διακόπτη η πρόεδρος. Κοιτάξτε, μιλάμε για την προσθήκη Απαιτήσει για ΦΠΑ υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος και για αυτή. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει έναν που ψηφίζει επιπλέον. Πέρα τη ψηφοφορία γίνεται δεκτό το επιπλέον αυτό τμήμα. We go to uh, amendment 31 uh, by 31. υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική Q αγγλικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική QA υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το QA. Υπάρχει πάντα ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρεστε στο QA. Υπάρχει και ένα DA. Αλλά το QA δεν υπάρχει. Το DA είναι αυτό που θα ψηφίσουμε τώρα. Το DA έρχεται μετά το QA, ε, λέει η Πρόεδρος. Μαρία δεν μπορούμε να κάνουμε εξαίρεση. Μπορείς να πας να φέρεις την κάρτα σου αν χρειάζεται ή κάποιος να στη φέρει. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την QA για μια ακόμη φορά. Ή μάλλον είναι ξεκάθαρο. Υπέρ 26-22 κατά. DA τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 41. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ή αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. M αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 59. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εξήντα. Προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Να αντικατασταθεί η λέξη η αγγλική fact από τη λέξη intention, πρόθεση, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή αλλαγή. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61. Δεκτή. «27 υπέρ 25 κατά». Συμβιβαστική H αγγλική υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική I. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική J. Επιπλέον τμήμα του κειμένου υπέρ. Θα σας διαβάσω τη φράση για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Υπενθυμίζει, <coughs> διακόπτει η Πρόεδρος εκ νέου, το H10. Αν γίνει δεκτή η συμβιβαστική J, το πρώτο τμήμα καταπίπτει και το δεύτερο είναι προσθήκη και λέει το κείμενο το εξή. Υπενθυμίζει τον έκτακτο χαρακτήρα των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, ιδιαίτερα τη πρόνοια και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και λέγεται ότι πρέπει να δοθούν εγγυήσει για την προσβασιμότητα ε, και την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 80 θα την πούμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30 κατά 23 υπέρ. 81. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΕΛΑ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 83. Πέρασε στις ψηφοφορίες 25 υπέρ, 23 κατά. 84 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική και υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 89 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ενενήντα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ενενήντα ένα έχει αποσυρθεί 91, συμβιβαστική M υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. «98 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή». «99 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή». «100 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή». Συμβιβαστική O υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική πι αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία υπαρίθμου 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή. Επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την επτά. ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 1. του α κεφαλαίου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, δεκτή, δεκτή, συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Στο β κεφαλαίο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το σύνολο τώρα της πρόταφης γνωμοδότησης όπως τροπολογήθηκε πέρας της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή 43 υπέρ, 8 κατά με τρεις αποχές. Έχει κανείς ε, αντίρρηση να το τοποθετήσουμε αυτό στα πρακτικά. Πολύ ωραία. Και το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη.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 Προχωρούμε λοιπόν όπως έλεγα στο σημείο 14 της ημισίας διατάξεω. γνωμοδότηση της Επιτροπή των Περιφερειών για τους μακροπρόθεσμα ανέργους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρώση, τον εισηγητή Τη Επιτροπή των Περιφερειών για να μας ε, κάνει μια δεκάλεπτη παρουσίαση εισαγωγή στην γνωμοδότηση αυτή για να έχουμε μετά ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, <clears throat> αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Vi ringrazio prima di tutto per questo invito a presentare il Σας παρουσιάζει λοιπόν την, ε, ε, την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών για την ένταξη των μακροπρόθεσμα ανέργων στην αγορά εργασίας. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω καταρχάς τη σημασία της δουλειάς που διεξέγεται από την Επιτροπή σας ε, επί σοβαρών κοινωνικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργασίας. Πρόκειται κατά την άποψή μου για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που απορρέουν από τη συνθήκη και οι οποίοι περιορίζουν, παρεμποδίζουν μια δεσμευτική ανάληψη δράσεως και πολιτικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών, εγώ εξέφρασα αποφασισμένα τη θέση αυτή, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να αντιμετωπιστεί αναγνωρίζοντας μια κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση που βασίζεται στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών που δεν θα πρέπει να αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικούν. Από εκεί και πέρα και από τα δεδομένα που έχουμε από την κοινωνική κατάσταση γενικώ τα ανησυχητικά δεδομένα που προκύπτουν την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, βλέπουμε ότι σήμερα ακόμα το 48,2% της συνολικής ανεργίας είναι μακροπρόθεσμη. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια μακροπρόθεσμα ανέργη. Μιλούμε δηλαδή για, τις, για ένα μέγεθος, μια διάσταση χώρας ολόκληρης. Το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να αποφασίσει, να το καταπιεί, να το τοποθετήσει στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω με την θέση του Συμβουλίου του Ιανουαρίου του 2016 που εξέφερσε ανησυχία για την ε, προκεχωρημένη πρόταση Κομισιόν να εισαγάγει ως δίκτυ εκτάκτου ανάγκης τον δίκτυ της μακροπρόθεσμης ανεργίας. η κοινωνική δείκτες και οι δείκτες επασχόλησης θεωρεί το Συμβούλιο ότι δεν είναι κατάλληλοι ώστε να εντοπιστούν μακροοικονομικοί κίνδυνοι. Αυτό είναι ένα λάθος κατά την άποψή μου. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσεως της χρηματοπιστωτικής κρίσεως θα έχει πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο της αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και της κοινωνίας. Η υποβάθμιση κοινωνική, η υποβάθμιση ακόμα και της υγείας. Οι κοινωνικές εντάσεις, οι πολιτικές εντάσεις προκύπτουν από την συνέχιση μιας κατάστασης <clears throat> δυσάρεστης, μιας μόνιμης κατάστασης μακροπρόθεσμης, όπως λέμε, ανεργίας, που αφορά σε 10 εκατομμύρια πολίτες. Και επ' αυτούς, επ του φαινομένου της μακροπρόθεσμης ανεργίας, θα ήθελα να πω ότι αν μη τι άλλο, εκφράζεται μια κάποια ευαισθησία ή ανησυχία προς το πρόβλημα, τονίζοντας την κεντρικότητα της σημασίας των υπηρεσιών απασχόλησης και εξέβρεσης της εργασίας. Αυτό όμως αφήνει ατόφιο το άχθος της προσπάθειας αυτής ένταξης στα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα στους δημόσιους φαρείς των κρατών μελών που πρέπει να δρουν χωρίς διακρίσεις. Οι υπηρεσίες λοιπόν ανεργίας που έχουν ήδη υποστεί πλήγματα από την κρίση θα πρέπει να αναλάβουν και αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν. Με μειωμένες επομένως πιθανότητες και αντιθέτως αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας αυτής της προσπάθειας. Ιδιαίτερα με τα, πιο, με αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Πρόκειται για μια περιοριστική, πολύ περιοριστική ερμηνεία της αρχής επικουρικότητας που δεν κάνει παρά να αποδυναμώνει. Να αποδυναμώνει την ήδη αποδυναμωμένη εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η Επιτροπή των Περιφερειών λοιπόν με ευρεία και οριζόντια αν θέλετε διαπολιτική πλειοψηφία ενέχρινε την γνωμοδότηση αυτή που λέει ότι πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις δεξιότητες και την κατάρτιση και αυτά θα πρέπει να τα ενσωματώσουν οι υπηρεσίες ενεργείας των κρατών μελών. Δεύτερον, θα πρέπει να καθορίσουμε δράσεις ευρωπαϊκές που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στα πρότυπα αυτά που θα έχουν καθοριστεί. Δεδομένων των τεράστιων αποκλήσεων και διαφορών που έχουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών και των δομών και των υπηρεσιών ανεργίας και της ίδιας της ενεργείας που διαφέρουν πάρα πολύ. Όλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν προς αξιολόγηση και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Τρίτον, οι διαρθρωτικές απαιτήσει του προβλήματος της ενεργείας, δηλαδή ότι το κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί δικού του πόρους ή πόρους που να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να γίνονται υπό πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση, σε σύγκριση με αυτές που προέρχονται από μια ευρύτατη και βαθύτατη κρίση επί του φαινομένου ε, επί του οποίου φαινομένου θα, μπορούσε να έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο αυξημένο, αν θέλετε, πιο ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο αντιμετώπισης. προκειμένου να αναλυφθούν αυτές οι προσπάθειες που είναι κοινή ωφελία, αν θέλετε, υπηρεσίες κοινού συμφέροντος και οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 14-20. Έτσι ώστε να ξεκινήσει επιτέλους μια συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων συζήτηση για το θέμα αυτό. Και πάντα στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής Κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο εγγυητικό μέσο για τους νέους. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε μια πρωτοβουλία για την μακροπρόθεσμη ενεργεία που πειραματικά εξετάσαμε στην δική μου περιφέρεια, στην Τοσκάνη. Δηλαδή, δημόσιοι διαγωνισμοί για την προσωρινή αποσχόληση εργαζομένων ιδιαίτερα ευάλωτων μακροπρόθεσμων ανέργων. Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση και από πλευράς των δημοσίων φορέων και από πλευράς ε, των ίδιων των ανέργων που ενδιαφέρθηκαν. Τώρα, πρέπει να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του τις συστάσεις και τις προτάσεις της ε, Επιτροπή των Περιφερειών και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε και των σχετικών παρατηρήσεων του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι οι πρωτοβουλίε πρέπει ακόμα πολλέ να αναλυθούν προ την κατεύθυνση αυτή, γιατί δεν έχει χαθεί η μάχη ακόμα. Και πρέπει να θυμίσουμε και την σημασία τη ανακοίνωση Κομισιόν για τη διαβούλευση σχετικά με τον αποκαλούμενο ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Λέγει η Κομισιόν ότι ο κίνδυνος μιας μακροοικονομικής κρίσης είναι κίνδυνος και απειλή για το σύνολο της Ευρωζώνης. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες αποκλήσεις τις αγορές εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες των κρατών μελών. Τι αξία έχουν τέτοιες δηλώσεις όμως αν δεν μεταφέρονται σε απτές και συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι θα είναι περιορισμένη η εξέτασή μας και η παρέμβασή μας αν δεν δούμε τη συνολικότερη εικόνα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της ενιαίας αγοράς εργασίας και να αποφύγουμε ενδεχομένως ο ασθενής κρίκος ή το ιδιαίτερο πρόβλημα του ενός κράτους να γίνεται πρόβλημα να μεταφέρεται και στο άλλο κράτος μέλος. Δεν θα ήταν καθόλου σοφό κάτι τέτοιο. Και δεν θα είναι δυνατό να οικοδομήσουμε μια ενιαία αγορά εργασίας σε χρόνους μηδέν, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε αν όλοι προσπαθήσουμε μαζί και δεσμευτούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρώση. Φυσικά ο αγώνας μας συνοδεύει με το δικό σας. Και δίνω το λόγο στους συναδέλφους που έχουν υποστηρίξει την υπόθεση αυτή από την Επιτροπή Απασχόλησης με την προφορική ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματος για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων. Ο κύριος Κάσα πρώτα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον κύριο Ρώση, πρώτα απ' όλα που ήρθε εδώ να μας μιλήσει και βέβαια για την εξαιρετική του παρουσίαση. Στη γνωμοδότησή της για την ένταξη των μακροπρόθεσμα ανέργων στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή των Περιφερειών αναφέρει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ιδιαίτερου ταμείου μιας εγγύησης για τους ενηλίκους, όπως τα λέγαμε, αντίστοιχης με την εγγύηση για την νεολαία, για τους μακροπρόθεσμα άνεργους. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει πιο πολλές λεπτομέρειες πώς βλέπει, από πού μπορούν να απορρέουν, δηλαδή τα κονδύλια για αυτό το ταμείο, ποιος θα μπορούσε να δικαιούται χρηματοδότηση από το ταμείο αυτό ή τι είδους συνέπειες θα μπορούσε να έχει ή αντίκτυπο για τους συμμετέχοντες. Έχει κάποια στοιχεία ο κύριος Ρώση να μας δώσει με πιο πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο κύριος Χαβιλόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τον κύριο Ρώση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και στο τελικό κείμενο που υιοθέτησε το Συμβούλιο. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές μετακινήσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε στο ψήφισμά μας στο Κοινοβούλιο ότι σε σχέση με αυτό το οποίο υιοθέτησε το Συμβούλιο, έχουν υπάρξει πάρα πολύ ουσιαστικές αλλαγές και να σας παρουσιάσω κάποιες από αυτές. Καταρχάς, η νομική βάση της συμφωνίας. Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως και η Επιτροπή, να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 149 του κανονισμού και τελικά χρησιμοποιείται το 148.2. Κάτι το οποίο ζητεί τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ως γνωμοδότηση και πέραν αυτού τίποτα. Εμείς ε, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όμως το συγκεκριμένο θέμα γιατί αφορά πολλά εκατομμύρια κόσμου και είναι σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το δικό μας ψήφισμα εξηγεί αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κατάλογο αυτό, το μητρό αυτό και λέμε ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις διοικήσεις των κρατών μελών αυτούς οι οποίοι είναι, μόνον αυτούς οι οποίοι είναι γεγραμμένοι, καταγεγραμμένοι. Τελικά το Συμβούλιο αποφασίζει ότι μόνο οι καταγεγραμμένοι θα λαμβάνονται υπόψη σε στατιστικό επίπεδο σαν α, μακροπρόθεσμα άνεργοι αντίθετα και από την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για την προσωπική αντιμετώπιση και τη χρονική προθεσμία. Εκεί το Συμβούλιο ε, θα έλεγα ότι ε, ποικίλει. Εμείς τονίζουμε ιδιαίτερα το ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρμοδιότητες και καθήκοντα ισορροπημένα και για τον ε, ενδιαφερόμενο και για την υπηρεσία εξέβρεση εργασίας. Το Συμβούλιο λοιπόν υποβάλλει μια πρόταση πάρα πολύ ανισόρροπη που τοποθετεί όλο το άκθος επί του εργαζομένου ή του ενδιαφερομένου. Και θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμό το άκθος που απορρέει από αυτήν την ανισόρροπη επαναλαμβάνω πρόταση του Συμβουλίου. Όμως θεσμικά αντιμετωπίζουμε την εξή κατάσταση. Η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση, έχει γίνει μια συζήτηση εδώ και κάποιους μήνες, εξετάζουμε και το συζητούμε το πράγμα και τελικά απέναντί μας τώρα βρίσκουμε μια πρόταση ουσιαστικά και θεμελιωδώς τροποποιημένη. Στην αρχή είχαμε συζητήσει για ένα πλαίσιο εργασίας και ότι θα είχαμε ένα εργαλείο για να αρχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα κτλ. Δηλαδή τελικώ η ερώτησή μου είναι τι θεωρείτε, τι πιστεύετε για αυτές τις ουσιαστικότατες, τις ριζικές τροποποιήσεις που υπέστη τελικώς αυτή η πρόταση. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις για να δώσετε μετά τις απαντήσεις σας. Ε, κυρία Σιγνάνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρώση για την παρουσίαση. Υποστηρίζω την ερώτηση του κυρίου Κάζα για το Ταμείο. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις της πτυχής αυτής. Ε, πόθεν θα τληθούν τα κονδύλια, ποιος θα τα δικαιούται. Και επίσης, με το παράδειγμα της Τοσκάνης, θα θέλατε να μας δώσετε για το παράδειγμα αυτό κάποιες ε, περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα των μακροχρόνιων έργων. Και βλέπουμε στη γνωμοδότηση Επιτροπής των Περιφερειών ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν και δημόσια δημόσιες προσπάθειες για την ένταξη των μακροχρόνιων έργων. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι εμείς στη Σλοβακία έχουμε νομοθεσία η οποία αναφέρεται βέβαια στη φτώχεια αλλά όταν γίνεται αυτή η παρέμβαση από το δημόσιο, ο μακρόνια ενεργός ε, δεν έχει κίνητρα να αναζητήσει μια θέση εργασίας και μάλλον καταχράται των δυνατοτήτων. Αντίστοιχα βλέπουμε μελέτες και από την Πολωνία, την Ουγγαρία. Έχετε κάποια παραδείγματα λοιπόν καλά, θετικά, όπου μπορεί να υποστηριχθεί αυτή η προσέγγιση από την πλευρά την κρατική. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω στον Ικαμιά και βλέπω ότι οι συνάδελφοί μου διερμηνείς είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και σας ευχαριστώ κύριε Ρώση για την ε, επισκόπηση. Δεν θέλω να σού υπερβολικά πολλές ερωτήσεις. Ήδη οι συνάδελφοι διατύπωσαν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, τις οποίες και υποστηρίζω. Είναι όντως πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Και φρονώ ότι δεν έχουμε αποδώσει αρκετή σημασία στο γεγονός ότι η μακροχρόνια ανεργή είναι τόσο πολύ εγκαταλελειμμένη από το σύστημα που ούτε καν μπορούμε να τους βρούμε, ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι. Και σε αυτό ευθύνονται βέβαια και οι τοπικές ε, ε, εκπρόσωποι, οι τοπικές αρχές. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να ασκηθεί η πίεση στα κράτη-μέλη και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην πατρίδα μου την Εσθονία όπου σε μία από τις ε, επαρχίες λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου κλείνουν εργοστάσια, μένουν άνεργοι πολλοί. Ζητούμε εμείς την κάλυψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης, από το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά ε, όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και με την ε, δημιουργία ενότητας συνεργασίας και τίποτα δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα λοιπόν πιο συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πώς μπορούμε να αποθήσουμε τα κράτη-μέλη στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδελφών επίσης ως προς το ποιος θα δικαιούται τα κονδύλια, ποιες διατυπώσεις θα προβλέπονται και βεβαίως πώς μπορούμε πάνω απ' όλα να τους επιτρέψουμε να επαναταχθούν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Λόπες Περνέιο. Ε, Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. 10 εκατομμύρια λοιπόν μακροπρόθεσμα άνεργοι. Πρόκειται για ένα μέγεθος ανυπόφορο. 10 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα. Ακριβώς αυτή, αυτό το μέγεθος είναι μια, ένα άμεσο αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας, μόνιμης λιτότητας, που έχουν εφαρμοστεί για τόσο καιρό. Επομένως, ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο θα είναι να απομακρυνθούμε επιτέλους από αυτές τις οικονομικές πολιτικές και τα μέτρα. Θα χρειαστεί ένα, μια πραγματική εφαρμογή πολιτικής ελάχιστου εισοδήματο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα στοιχεία κοινωνικής προστασίας, τις κοινωνικές παροχές ανεργίας, τα επιδόματα, τα οποία έχουν εγκαταλείψει οι αρχές, οι χώρες με συγχωρείτε. Και μαζί με αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να αναπτύξουμε ενεργείες πολιτικές απασχόλησης για την απασχόληση για την αγορά εργασίας και αυτό θα πρέπει να σχετίζεται όχι μόνο με τις επιχειρήσεις αλλά με ένα συνολικότερο πρότυπο παραγωγικό που να καταλήξει σε ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Ε, εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο και αυτό το αναφέρει και το ελεγκτικό συνέδριο ότι ο περιορισμός των επιδομάτων όπως συνέβη στα πλαίσια των ε, εγγυητικών μέσων για την νεολαία δεν λειτουργήσαν και δεν έδωσαν τα αποτελέσματα που ελπίζαμε ότι θα έδιναν. Δεν μπορούμε να συνδέουμε τα πάντα με προσωρινές συμβάσεις εργασίας εθελοντικές. Δεν ταυτίζεται καθόλου αυτό με τις ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης που επιθυμούμε. Ούτε η μείωση των εισφορών. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και αυτό να το κάνουμε μαζί με τους κοινωνικούς φορείς και η Κομισιόν θα πρέπει να στοιχηματίσει στην εργασία, να επενδύσει στην εργασία. Δηλαδή θα πρέπει να ασχολούμαστε λιγότερο με τα χρηματοπιστωτικά πράγματα και περισσότερο με το να έχουμε ένα παραγωγικό πρότυπο, πρότυπο καινοτόμο που να καταλήγει σε βιώσιμη απασχόληση. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν είστε εδώ. Δεν είμαι. Η κυρία Ράγκε, βέβαια στο σύνομαι εκ μέρους της και την αντικαθιστώ. Θέλει να σημαίνει τις εξής ε, σκέψεις μέσα καθώς έχει μελετήσει το θέμα. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξή. Πρέπει να εξασφαλιστεί υποστήριξη εισοδήματο, στήριξη εισοδήματο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη αρνητική εκκίνηση και τη αιρεσιμότητα. Πρέπει να στηριχθούμε στη βοήθεια των οργανώσεων εκείνων που έχουν μακρά εμπειρία από την ένταξη στην αγορά εργασία των ε, μακροχρόνιων ενέργων. Εμεί, οι πράσινοι δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο σε εκστρατείε ευαισθητοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένους πόρους για το συγκεκριμένο έργο. Ε, δεν θα πρέπει να προσδιορίζεται στην ε, ατομική αξιολόγηση μόνο η απασχολησιμότητα και η πορεία μιας σταδιοδρομίας, αλλά θα πρέπει σε αυτή να περιλαμβάνονται μια αξιολόγηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον μακροχρόνια άνεργο και διευκόλυνση για την αντιμετώπιση των προσκομμάτων που θα βρει στην πορεία του. Επίσης, καλωσορίζουμε μέτρα για μια πιο ανοιχτή προς όλους ε, αγορά εργασίας, μέτρα δηλαδή τα οποία θα βοηθήσουν στην ένταξη στην αγορά. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε και πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη ακόμη. Γι' αυτό προσπαθήστε παρακαλώ να είστε συνοπτικοί και να μην επαναλαμβάνετε αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Ατζία. Να καλωσορίσω και εγώ τον Πρόεδρο κύριο Ρώση. Πραγματικά η αίσθηση της ομιλίας σας εκφράζει θα έλεγα τη θλίψη της μετά τον θάνατο συγκεκριμένου προσώπου πολύ γνωστού και τον τραυματισμό δύο άλλων. Είναι σαφές ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν κινδύνους και ακόμα και στη Τοσκάνη απαιτούνται ε, προσπάθειες ε, ιδιαίτερα για την ε, επικίνδυνες εργασίες. Δεν αρκεί ένα κράνος για να προστατευτεί η ζωή αυτών οι οποίοι εργάζονται κάτω από το έδαφος πολλές φορές και δυστυχώς οι συνθήκες εργασίας σε περιοχές όπως τα ορυχεία της Καράρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και το μόνο που κάνουν είναι να βοηθούν τις πολυεθνικές να κερδίζουν περισσότερα. Η δική σας περιοχή συνδέεται με την Ευρώπη και πρέπει να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με την Ευρώπη. Χάρη ακριβώς και στους συναδέλφους της περιφέρειας της Τοσκάνης, και τους εκπροσώπους της περιφέρειας αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καταθέσει σαν παράδειγμα ερωτήσεις παφορικές για τα γκάλα, τις τοπικές ομάδες πρωτοβουλίας που κανονικά θα έπρεπε να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να βοηθούν τους νέους να βρουν δουλειά, να εμποδίζουν τον κόσμο ουσιαστικά να φεύγει από την περιοχή. Και όμως αυτά τα γκάλα δυστυχώς οδήγησαν στην απώλεια εκατομμυρίων ευρώ. Πώς μπορεί λοιπόν οι ιδέες να είναι καλές και στην πραγματικότητα να διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση στις περιφερειές μας είναι εντελώς διαφορετικής και αναφέρομαι και, στον γκάλ, και σε συγκεκριμένα γκάλ της Τοσκάνης, όπως την Καφάνια κτλ. Νομίζω ότι ε, είναι μια απλή ερώτηση αυτή την οποία ε, έκανα. Δεν ε, περιμένω βέβαια να απαντήσετε όπως ο Παντοάν, ο οποίος όταν του θέτουν ερωτήσεις για την Ιταλία δεν δίνει ποτέ απαντήσεις. Ποιες είναι οι ευθύνες λοιπόν για την περίπτωση της τράπεζας Monte dei Paschi και οι σχέσεις της με την περιφέρεια της Τοσκάνης γενικότερα. Δώστε μου παρακαλώ κάποιες απαντήσεις. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί μου το ζητήσατε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο επιλογές οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Ένα τμήμα, θα έλεγα όπως η Εστονία εκπρόσωπος, είπε ότι δεν χρειάζεται να επιδοτούμε τους ανέργους, μόνο να τους δώσουμε δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια δουλειά. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσουν τα αίτια. Και νομίζω ότι εδώ πραγματοποιούμε σημαντική πρόοδο αν τα καταφέρουμε. Στα αίτια δηλαδή της μακροχρόνιας ενεργείας. Η παγκοσμιοποίηση την οποία εσείς επιθυμείτε και υποστηρίζετε είναι ένας από τους πραγματικούς λόγους. Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών. Και πάλι σήμερα είδαμε με την, με την Κορέα, ε, με το TTIP, την Κίνα. Βλέπουμε ότι αυτά τα διαδοχικά ανοίγματα των αγορών έχουν σαν αποτέλεσμα οι χώρες low cost να ωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση. Και το κοινωνικό dumping αναπτύσσει πλήρως τις συνέπειες του, γεννώντας μακροχρόνια άνεργους. Έχετε νομίζω εξουδετερώσει κάθε τελωνιακή προστασία και όταν καταργούνται οι τελωνιακές προστασίες φτάνουμε σε διεθνείς ε, κατακλυσμούς εις βάρος των εργαζομένων. Ε, και ο, καθώς θέλετε να διανύμετε ε, ε εισόδημα στους πάντες, καταργείτε εν τέλει την υποστήριξη προς τον φτωχό. Η κατανομή αυτή του πλούτου φτωχαίνει τον κόσμο. Είναι σαν να κόβεται κομματάκια την κότα με το χρυσό αυγό. δεν υπάρχει τίποτα να μοιραστεί στους φτωχούς. Ε, Ευχαριστώ. Μπενεφάι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Ενρίκο Ρώση, τον πρόεδρο Ρώση, είναι πάντα θετικό το να μπορεί κανείς να συνομιλήσει με τον πρόεδρο μιας τόσο σημαντικής ευρωπαϊκής περιφέρειας, η οποία έχει καινοτομήσει τα μάλα, με πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμη φορά όμως την ανησυχία μου για το φαινόμενο της ανεργίας της μακροπρόθεσμης που είναι σε ανησυχητικά επίπεδα το είμαι ικανοποιημένος τώρα και από την ικανότητα που έχει η Επιτροπή των Περιφερειών να εντοπίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της συζήτησης και να αναζητεί φιλόδοξες λύσεις. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ουσιαστικές, ανάγκη ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα πρέπει να βελτιωθεί επίσης η εγγύηση για τους νέους στο μέσο αυτό και θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία και με βάση τις προτάσεις τις οποίες μας παρουσίασε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή ο Υπουργός Παντοάν. Τώρα και το Συμβούλιο, όπως είπε ο κύριος Χάβη Λόπες, έχει προβλέψει ένα νομικό μέσο το οποίο είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει βέβαια να προσπαθήσουμε εμείς να προωθήσουμε την πλατφόρμα αυτή που περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα, τα ποιοτικά, γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών δίνει την δυνατότητα υπηρεσιών οι οποίες είναι κατάλληλες γιατί λαμβάνουν υπόψη τις επιτόπου ανάγκες και βελτιώνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων σε μια αγορά εργασίας η οποία βρίσκεται σε μόνιμη αλλαγή. Τα κέντρα για την απασχόληση στην Ιταλία δυστυχώς όμως για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα σημείο αδυ, αδυναμίας και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν πραγματικά τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν αντίθετα από χώρες όπως η Γερμανία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξουν αλλαγές και στην χώρα μου γύρω από αυτό, να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός επίσης των διαδικασιών για την απασχόληση και στα πλαίσια της εγγύησης για τους νέους και αυτό φάνηκε και στην τελευταία έκθεσή μας ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις βέλτιστες πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε εκεί που χρειάζεται. Κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία παρά τις κριτικές και μπορεί να αποδώσει εφόσον βέβαια οι πρωτοβουλίες συνδυαστούν σωστά με τα υπάρχοντα μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας, την βελτίωση της απασχολησιμότητας και ε, μέτρα υπέρ της απασχόλησης των νέων. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον κύριο Ρώση και περιμένω την άποψή του. Ε, δεν θα ήθελα η συζήτηση να γίνει σε αυστηρά εθνικό επίπεδο γιατί αυτό ίσως να μην ενδιαφέρει κάποιον άλλο εδώ. Τόμας Μαν. Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχουν ως καθήκον να αναζητούν συμβαστικές ε, λύσεις και μπράβο τους, αυτό μπορούν να το καταφέρουν σε πολλούς τομείς, εμείς όχι πάντα βέβαια. Εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με την παρουσίαση μιας τελικής περιφερεια λιγότερο με την Ευρώπη και θέλω και σε αυτό να συμφωνήσω με τον συνάδελφο γιατί θα ήταν πιο σημαντικό νομίζω να είναι ορατότερη η ευρωπαϊκή διάσταση και όταν ε, Βλέπουμε βεβαίως ε, αυτό το επαναλαμβανόμενο ότι όλα καταστρέφονται κτλ. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις, σε παραδείγματι με στοχευμένη διαθέση των κονδυλίων στη Γερμανία, επί μέσα στην κρίση δεν ε, ε, καταβάλλονταν ε, επιδόματα ενεργείας αν υπήρχε διαθέσιμη για τον ανεργοθέση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας κύριε Ρώση, ώστε να μην αφήσουμε στους ε, ακραίους της δεξιάς επιχειρήματα πρέπει να μην αφήσουμε να μετακυληθεί η επιχειρηματολογία προς το θέμα των προσφύγων και να γίνουν οι επενδύσεις εκεί που χρειάζονται και βέβαια εδώ έχουμε την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ενεργείας και είναι πολύ σωστή η επιλογή του θέματος. Πολύ σωστά λέτε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν υλοποιούνται ή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν μέτρα περιφερειακά και αναπτύσσονται, το βλέπω και εγώ στη δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα, με, ε, με υποστήριξη από το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά εάν δεν υπάρχει αυτό, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κέντρα καταπολέμησης της φτώχειας, όπου τα κράτη-μέλη λένε «Α, όχι, θα τα καταφέρω μόνος μου», αλλά μόνο το κάθε κράτος δεν μπορεί να το ε, επιτύχει αυτό. Πρέπει να καταστήσουμε απόλυτο σαφές ότι υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και πρέπει να καταστεί ορατή η προσθέμενη αξία και να προβάλλεται πάντοτε. Γι' αυτό λοιπόν στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει πιστεύω στην ε, γνωμοδότηση σας να ε, εντοπιστούν και να συνδυαστούν με συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να καθίσετε ορατό ότι εμείς ως Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και επιτυγχάνουμε πολλά πράγματα για την καταπολέμηση μικροχρόνιας ενεργείας. Είναι πολύ καλή, πολύ εύστοχη η γνωμοδότηση σας, αρκεί να προχωρήσουμε με αποτελεσματικότητα και στους δύο τομείς για να κερδίσουμε και την αποδοχή της Ευρώπης από τον πολίτη, ώστε να μην αφήσουμε επιχειρηματολογία για τους ακραίους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάσου Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Ρώση, για την εμπειρία από την προσωπική σας εμπειρία που μας ε, αναφέρατε. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει συνδετικός κρίκος μεταξύ ε, κατάρτισης και απασχολησιμότητας και μάλιστα για αυτό το λόγο πήγα, πήρα το λόγο γιατί έκανε αυτή την παρατήρηση συνάδελφος. Εγώ από την Πολωνία έχω συγκεκριμένα πολύ καλά αποτελέσματα καταγράψει από αυτή την προσπάθεια. Πολύ συχνά ακούγονται διαμαρτυρίες, ε, ειδικά τελευταία, ότι δεν ε, εξοπλίζει το μορφωτικό, το εκπαιδευτικό σύστημα το νέο ώστε να μπορέσει να μπει σε μια σταδιοδρομία, ώστε να έχει τα προσόντα που χρειάζεται για την ε, ένταξη στην αγορά εργασίας. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε με την ε, κατάρτιση, την περαιτέρω διαβίου μάθηση, να υποστηρίξουμε το νέο για να αποκτήσει τις περαιτέρω δεξιότητες που χρειάζεται μετά το σχολείο. Και νομίζω ότι η κατάρτιση θα πρέπει να επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες και προετοιμασία. Πρέπει να γίνει βεβαίως η ανάλυση των αναγκών και να εξευρεθούν οι εκπαιδευτές εκείνοι οι οποίοι θα συμπληρώσουν τις ελλείψεις σε δεξιότητες και άλλα προσόντα. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι πολύ συχνά στην Επιτροπή μας απευθύνω έκκληση για την συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ξεκινώντας από το περιφερειακό κυρίως, για την αγορά εργασίας ιδιαίτερως. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει η ανάλυση των δεδομένων και αντίστοιχα η αναζήτηση των λύσεων όταν στη διάθεσή μας έχουμε μόνο συμπιλημένα εθνικά ε, στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν δείχνουν ξεκάθαρα την ε, πραγματικότητα. Μιλούμε για δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, που δεν έχουν καλυφθεί ενώ υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων ανεργοί που δεν μπορούν να έχουν ε, την επαρκή κατάρτιση που θα τους επιτρέψει να αναλάβουν τις δεξιότητες για να καλύψουν τις θέσεις αυτές και δεν έχουν και κανένα να τους καθοδηγήσει. Γι' αυτό λοιπόν η συλλογή των δεδομένων σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χρήσιμη πιστεύω. Θέλω τη δική σας θέση, καθώς βέβαια και τις θέσεις σε σχέση με την κατάρτιση. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη κατάρτιση νέου. Thank Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρουσιάσεις σας. πολλές ερωτήσεις. Δεν πρέπει μόνο να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις μόνο, αλλά πρέπει να μεταφέρετε και το δικό σας μήνυμα. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και για το πάθος το οποίο επιδεικνύεται για τα θέματα αυτά και το οποίο συμμερίζομαι θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Ατζέα, η οποία με ανεπίκαιρο τρόπο μου θέτει πάρα πολλές ερωτήσεις για το σύνολο των ευρωπαϊκών περιοχών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα απαντήσω στην κυρία Ατζέα με ευγένεια και γραπτά, ζητώντας της ίσως να αναγνώσει την απάντησή μου στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής σας, στην οποία δεν μετέχω. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να πω ότι σχετικά με τα γκάλ, εμείς πάντα θεωρήσαμε ότι ήταν μια σωστή πρακτική ε, και αυτό είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωση της Τοσκάνης, αυτό το οικονομικό Ινστιτούτο στο οποίο συμμετέχει η περιφέρεια. Αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες λοιπόν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα για να βοηθήσει ένα δις 400 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια προς τους βιοτέχνες της περιοχής. Σχετικά με το θέμα των Απουάνε που είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό είναι μία από τις λίγες περιφέρειες στην Ιταλία, εμείς και η Απουλία το κάνουμε αυτό, φροντίδας του φυσικού κάλου της περιοχής και του φυσικού ταπείου οποίο, συγγνώμη, και σε σχέση με τις ανασκαφές. Και έχουμε περάσει ένα νόμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ε, περάσει σε επίπεδο εθνικό, που υποχρεώζει αυτούς που αναλαμβάνουν τις ανασκαφές ε, να χρησιμοποιήσουν περισσότερο κόσμο από ό,τι γίνεται σήμερα. Και ιδιαίτερα για την περίπτωση των ε, ορυχείων μαρμάρου των λατομείων μαρμάρου που παρέχουν πάρα πολλά κέρδη και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και ιδιαίτερα θα πρέπει να κλείσουν οι σύραγγες στις οποίες υπάρχουν και γίνονται σοβαρά ατυχήματα που οφείλονται ακριβώς στον μη σεβασμό των βασικών κανόνων ασφαλείας. Θα απαντήσω αναλυτικότερα λοιπόν σε σχέση με όλα αυτά. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να πω βλέποντας και γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό σύστημα και πώς λειτουργεί νομικά το σύστημα αυτό για την ευρωπαϊκή παρέμβαση, είναι ότι μου ζητήθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών μου ζήτησε να προετοιμάσω αυτή τη γνωμοδότηση και στην αρχή νόμιζα ότι είχα να κάνω με κάτι το καινούριο όπως ακριβώς το έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη είναι κάτι το οποίο ε, εξελίσσεται μόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν γίνεται γι' αυτό συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα αλλάζουμε το παιχνίδι και αυτό το οποίο βγαίνει και από πλευράς του Συμβουλίου, αυτό το οποίο προτείνεται τώρα, Επαναλαμβάνω ότι ήδη το δικό μας ψήφισμα είναι καρπός συμβιβασμού, όπως και είχε υπογραμμίσει και ο κύριος Τόμας Μαν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώθηκε η εμβέλεια των προτάσεων τις οποίες είχαμε κάνει και φοβάμαι ότι η Ευρώπη στον τομέα αυτό δεν έχει αναπτυχθεί πολιτικά όσο χρειάζεται για να παρέμβει. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επί της ουσίας αντιπαραθέσεις. Από τη μία υπάρχουν χώροι παρέμβασης, από την άλλη υπάρχουν δυνατότητες για τον περιορισμό. 151 και 153 των συνθήκων δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω τα άρθρα αυτά, μπορεί και να τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Η διέξοδος την οποία εμείς αναζητήσαμε είναι να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη μορφή ανεργίας την οποία θα χαρακτηρίζαμε διαρθρωτική. Εγώ με την έννοια αυτή δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος, αλλά όπως είπα η πρότασή μας είναι καρπός συμβιβασμού. Μιλάμε λοιπόν για μια διαρθρωτική απασχόληση. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για πλήρη απασχόληση, κάτι το οποίο όμως δημιουργεί προβλήματα πολιτικά. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλοι μιλούσαμε για την πλήρη απασχόληση. Τώρα δεν μπορούμε να το προωθήσουμε ούτε καν σαν μια ιδέα επιμέρους και φαίνεται ότι είναι πολύ εκρηκτική, πάρα πολύ ριζοσπαστική και μιλάμε μόνο για μια διαφθρωτική μορφή ανεργίας σε διάφορες χώρες ε, όπου απαιτείται μια δυνατότητα ευρωπαϊκής παρέμβασης με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της απλής αρχής των επικοινωνούντων δοχείων και τα διάφορα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ένωση προσπαθούν να κατευνάσουν τις κοινωνικές εντάσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεργία με μέτρα όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμείς προτείνουμε το εξή, αν και εμένα δεν μου αρκεί προσωπικά, αλλά προτείνουμε την έννοια αυτή της ανεργίας της διαφθορτικής με την οποία πρέπει να ασχοληθούν οι κυβερνήσεις και μετά μια άλλη μορφή ανεργίας ε, με την οποία θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί περισσότερη έρευνα, περισσότερη ανάλυση, περισσότερες συζητήσεις και σε πιο τεχνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο που παίζουν τα κέντρα για την απασχόληση. Από χώρα σε χώρα σε σχέση με τα κέντρα αυτά απασχόλησης οι διαφορές είναι τεράστιες. Εγώ είμαι πρόεδρος μιας περιοχής και μιας περιφερειακής επιτροπής που ασχολείται με τις σχέσεις με την κεντρική κυβέρνηση να σχολιάσω τα προγράμματα για την απασχόληση στην Ιταλία και αναφέρθηκε σε αυτά και ο κύριος Μπονιφέη. Έγιναν κάποια θετικά βήματα, αλλά σε σχέση με την Γερμανία σαν παράδειγμα οι διαφορές μας είναι τεράστιες. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα βέβαια στην Ιταλία αλλά το σύνολο των εργαζομένων στην Ιταλία ε, εργάζονται στα κέντρα αυτά 3.000 ε, υπάλληλοι, ενώ στην Γερμανία 30.000. Ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στον πληθυσμό των δύο χωρών, καταλαβαίνετε ότι το κράτος παρεμβαίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ ε, σωστό, σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Λοιπόν, για τους νέους, δεν είναι αλήθεια αυτά που, διαβάνετε, που διαβάζετε στις εφημερίδες. Ε, εμείς με τα μέτρα που πήραμε καταφέραμε στην Ιταλία παρά την έλλειψη του προσωπικού των κέντρων απασχόλησης να βοηθήσουμε δεκάδες χιλιάδες νέους των οποίων γνωρίζουμε πια τις αντιλήψεις, τις δεξιότητες, τις διαθεσιμότητες και το τι μπορούν να προσφέρουν. Λοιπόν, ας ενισχύσουμε τα κέντρα για την απασχόληση. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να είναι αντίστοιχα, ομόλογα με το αίτημα για εργασία, με την ζήτηση που υπάρχει για θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους ανέργους, ιδιαίτερα τους μακροπρόθεσμα ανέργους, και να είναι πιο σωστά προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στην ζήτηση για θέσεις που αναπτύσσουν στον ιδιωτικό τομέα οι επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν βασικό εδώ το θέμα της πληροφόρησης. Εγώ έχω ε, πάρα πολλές επαφές με τους εργοδότες, με τους επιχειρηματίες και το να έχει κανείς μια σωστή επαγγελματική κατάρτιση και να μπορεί να προσφέρει εργαζομένους οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις παραγωγικές ανάγκες, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι βασικό για τον επιχειρηματία, είναι βασικό για τον εργοδότη. Είναι σαφές και αποδεδειγμένο πλέον ότι το ανθρώπινο δυναμικό σωστά καταρτισμένο είναι βασικό όπλο για την ανάπτυξη μιας χώρας. Συνεπώς λοιπόν το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να συνδέσουμε τα κέντρα για την απασχόληση με τις γνώσεις και την κατάρτιση για τις ανάγκες της εργασίας, να έχουμε σωστά profiling για τους εργαζομένους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα διάφορα κέντρα και όλα αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή η προσφορά με τη ζήτηση. Τώρα, σχετικά με τα κέντρα απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Αν και τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή διευκρινιστεί η μορφή της διαφθορτικής ανεργίας, θα παρέμβουν με το δικό τους τρόπο. Εγώ θα έλεγα ελπίζω έτσι ώστε η Ευρώπη να δώσει κάποια κίνητρα για τα κέντρα αυτά για την απασχόληση να μας πει ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν και να παρέχονται προς τους ανέργους και τις οποίες μπορούν να βρίσκουν ακριβώς τα κέντρα για την απασχόληση που είπα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στον τομέα της εργασίας και που προετοιμάζει ακριβώς την προσφορά στην ζήτηση. Αν καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πετύχουμε, να το πετύχουμε, αυτό θα είναι βασικό. Έχουμε χρόνο, απαιτείται χρόνος μάλλον, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ας έχουμε τον κατάλληλο χρόνο για να το πετύχουμε. Τέλος, πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε και με ένα πρόβλημα οικονομικό. Νομίζω ότι έχουμε μια κάποια ευκαιρία βέβαια, μια μεγάλη ευκαιρία να παρέμβουμε ξανά για το θέμα όταν συζητήσουμε το θέμα της επανεξέτασης, της ανακατανομής των ταμείων στην προγραμματική περίοδο 14-20. Η ενδιάμεση αξιολόγηση θα γίνει τον επόμενο χρόνο και οι συζητήσεις ήδη ξεκίνησαν. Οι δυνατότητες παρέμβασής μας μπορεί να είναι διπλές. Από τη μία αύξηση των διαθεσίμων ποσών. Έτσι να διευκολύνουμε κατά κάποιο τρόπο την ζήτηση, αν θέλετε, κάτι το οποίο έχει ανάγκη η Ευρώπη. Εμείς ελπίζαμε να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό πιστεύαμε ότι ήταν στοιχείο δικαιοσύνης, όχι μόνο οικονομικό στοιχείο. Εγώ δεν θέλω να ασκήσω οποιαδήποτε μορφή πολεμικής, αλλά βλέπω με εντύπωση περίεργη όταν επιλέγουν την εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων οι χώρες και όταν πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα γι' αυτό διστάζουν. Λοιπόν, ε, δεν μιλάμε για δις εδώ. Νομίζω ότι το θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας είναι κάτι το οποίο έχουμε αγνοήσει εν πολλής ε, σαν ευρωπαϊκά όργανα και αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο τα ευρωπαϊκά όργανα κινδυνεύουν να απολέσουν αξιοπιστία, να απολέσουν αυτό το στοιχείο εμπιστοσύνης το οποίο πρέπει να τρέφουν απέναντί τους οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και από την άλλη θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και να καταλήξουμε σε νέες ευελιξίες, ειδικά στις χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας και τις περιφέρειες που έχουν ε, τέτοια επίπεδα. Εμείς έχουμε, και το λέω αυτό, χωρίς να έχω προσωπικό συμφέρον, η περιοχή της Τοσκάνης έχει επίπεδα ανεργίας πολύ χαμηλότερα από το μέσον όρο της χώρας μου. Σας ευχαριστούμε <clears throat> κύριε Ρώση που μοιραστήκατε μαζί μας όλα αυτά τα στοιχεία και, όλοι και όλες αυτές τις ιδέες και τοποθετήσεις. Αυτή εδώ η Επιτροπή ακριβώς αυτά τα θέματα εξετάζει και συζητά. Και ακριβώς αντίστοιχες με τις δικές σας είναι και οι δικές μας στοχεύσεις. Ώστε σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης να έχει κανείς τη δυνατότητα να εργάζεται και να εξελίσσει τον εαυτό του. Πριν από λίγους μήνες εγκρίναμε ε, μία έκθεση της Επιτροπής αυτής σχετικά με υπηρεσίες απασχόλησης, ένα νέο είδος έουρες, δηλαδή μια διασύνδεση όλων των μέσων, όλων των υπηρεσιών και των φορέων των διαφόρων κρατών μελών, που να βοηθούν τους Ευρωπαίους πολίτες παντού και στην Ήπεθρο και εκτός των αστικών κέντρων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά δεν είχαν τελικώ χρόνο να πάρουν το λόγο σήμερα, αλλά θα τα συνασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, λέει η πρόεδρο. μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της μισής διατάξεως, που είναι το 15. το δυνητικό δημιουργία θέσεων απασχόληση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Κρασνοντέψκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει και το επόμενο σημείο της διατάξεως. Αυτό εδώ δηλαδή με ένα ίδιο ζήτημα, ένα ίδιο πρόβλημα υπό μια άλλη οπτική γωνία. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση από πλευρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια ομάδα των επιχειρήσεων που συνεχώς επαναλαμβάνουμε την αξία της και τη σημασία της στις τοποθετήσεις μας στο Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν όμως των δηλώσεων και των τοποθετήσεων και της αναγνώρισης που γίνεται προς τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές σημαντικότατα προβλήματα. Εγώ προσπάθησα λοιπόν στην γνωμοδότησή μου να απαριθμίσω κάποια από τα προβλήματα αυτά, ίσως όχι όλα, προσέγγισα το θέμα επιλεκτικά, ώστε να υπογραμμίσω τα πιο σημαντικά θέματα. Μερικά από αυτά είναι η φυγή εγκεφάλων, η έλλειψη εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες και κατάρτιση, και βεβαίως ο ρόλος και το ειδικό βάρος των πολυεθνικών, των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Προσπάθησα να ακολουθήσω μία δομή σαφή και ανοιχτή σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με τη δημιουργία εργασίας εστιαζόμενος σε συγκεκριμένα φαινόμενα και διαδικασίες τα οποία, στα οποία αναφερόμαστε συχνά αλλά ίσως όχι με παρκώς λεπτομερή τρόπο ή περιγραφικό τρόπο. Σχετικά με μια τάση πιο ακαδημαϊκής αν θέλετε τοποθέτησης ή άποψης για κάποια επαγγέλματα που είναι φαινόμενα που τελικώς αποθαρρύνουν τις μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το να αν προσλαμβάνουν νέους εργαζομένους, από το να δημιουργούν δηλαδή θέσεις απασχόλησης. Και θα έπρεπε να σκεφτούμε και οικονομικά, χρηματοδοτικά κίνητρα για την απασχόληση των νέων. Γιατί το να εργάζεται κανεί σε μια μικρή επιχείρηση δεν είναι πάντοτε αναγκαστικά μια ελκυστική, δεν θεωρείται αναγκαστικά μια ελκυστική θέση απασχόληση. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση για τα προγράμματα κατάρτιση στα πλαίσια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τα προγράμματα άσκησης και χρειάζεται επίσης μια ενθάρρυνση και μια ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Αυτά είναι στο πρώτο τμήμα της ε, γνωμοδότησης. Το δεύτερο τμήμα αφιερώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο, αν θέλετε. Σε επαφές, σε πολλές επαφές που είχαμε εκπροσώπους των επιχειρήσεων, λένε όχι μόνο ότι είναι υπερβολικά περιοριστική η νομοθεσία, αλλά ότι σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει ασάφεια στην νομοθεσία και υπάρχει και συνεχής τροποποίηση, εναλλαγή, ένα ρευστό νομικό πλαίσιο. Και κυρίως όλες αυτές οι διατάξεις που υπάρχουν, υπάρχουν πάνω απ' όλα ώστε να, στα απολύτως στα μέτρα των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και ώστε να υποστηρίζουν εκείνες. Επομένως, αν θέλετε, το νομικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ακριβώς το αντίθετο. Στο τελευταίο μέμα της ε, γνωμοδότησης ασχολούμαι με τον δίκαιο ανταγωνισμό. Το έχουμε ακούσει και σε άλλες συζητήσεις, σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Είναι κοινό τόπος ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν δυσμενέστερη αντιμετώπιση φορολογική από τις άλλες επιχειρήσεις. Το είπε πρόσφατα και ο Επίτροπος, ότι δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλύτερο φορολογικό άχθος κατά 30% επί των ΜΜΕ. Και αυτό λόγω της οικονομίας κλίμακος ή και της φοροδιαφυγής που ακολουθείται συστηματικά από τους πολύ μεγάλους ομίλους. Ακούσαμε και διαβάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στις τελευταίες αποκαλύψεις των Panama Papers και τα λοιπά. Το πρόβλημα πάντως της ανταγωνιστικότητας είναι και ένα πρόβλημα δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής στο νομικό πλαίσιο παρότι επαναλαμβάνω ότι αυτό το νομικό πλαίσιο είναι εποφελέστερο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο τρίτο τμήμα της νομοδότησης αναφέρω και ένα άλλο στοιχείο που το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα ήθελα να καταστεί προφανές ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι, έχουν πολύ ισχυρότερη παρουσία σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, σε κάποιες χώρες από ότι σε κάποιες άλλες. Επί τα νεότερα, τα πιο πρόσφατα κράτη-μέλη. Οικοδόμησαν την οικονομία τους της ελεύθερης αγοράς μετά το 1990 και στην ουσία εισάγοντας απλόχερα πολυεθνικές και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στο έδαφος τους για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις και εν τέλει άλλη ρυθμιστική και νομοθετική αντιμετώπιση. Αυτό είναι απολύτως εμφανές και είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αυτή η διαφοροποίηση δηλαδή που υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλούμε για ένα ισότιμο παιχνίδι και έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Διότι στο τέλος οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως συχνά λέμε είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και αντιπροσωπεύουν και την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του επιχειρήν σε μεγέθη. Είχα κάποιες πρώτες ανταλλαγές με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία ώστε αυτή η γνωμοδότηση να μπορέσει ακόμα περισσότερο να βελτιωθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα έγγραφο, μια έκθεση που θα μπορεί να έχει τουλάχιστον μια σαφήνεια και επιτυχία γιατί ο τελικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να καταπολεμήσουμε, να περιορίσουμε τη μάστιγα της ενεργείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο πρόεδρος, ο Ντέιβιντ. Αναλαμβάνει ο κύριος Μπαχ. Καλώς ευχαριστώ. Θα σας ε, διαβάσω την, τις παρατηρήσεις κυρίας Κλούνια και δεν μπορούσε να έρθει η ίδια σήμερα για να τις παρουσιάσει. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή του δουλειά, για την έκθεση, η οποία καλύπτει μια σειρά από τομείς και θέματα που πιστεύω έχουν μεγάλη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εστιάζεται λοιπόν η, η έκθεση στην πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση, τις δεξιότητες, ένα ισότιμο φορολογικό σύστημα, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα κέρια ζητήματα. Ως εκπρόσωπος βέβαια του ΕΛΚ και σκιώδης συγκέντρια πιστεύω ότι πρέπει να προσταθούν κάποια σημεία ακόμη στην έκθεση σε σχέση με, το, με τα προβλήματα ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της, ε, του συγκερασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες για διευθετήσεις ε, και κίνητρα έτσι ώστε να μπορεί κανείς να δουλεύει με καλύτερες συνθήκες και να εργάζεται περισσότερο. Επίσης, ιδιαίτερη μέρη να πρέπει να ληφθεί για τους ε, γονείς που μόνοι τους ανατρέφουν τέκνα και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και τη σχετική φορολογία, ε, την δυνατότητα να αναπτυχθούν ε, νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα πρέπει να απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκκληση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, κανονιστικό, ώστε να διευκολύνεται το crowdfunding και η επένδυση σε αγορές χάρη σε crowdfunding σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επεξεργάζονται τη δημιουργία μονοθερητικής ε, προσέγγισης για κάθε κανονιστική απέτηση, κάθε νομοθετική απέτηση. Αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας. Ε, τέλει, και σε σχέση με την ε, εκπαίδευση πρέπει να αναλυφθούν μέτρα προκειμένου να αναγνωριστούν οι δεξιότητες και τα προσόντα, διπλώματα και άλλα ε, πιστοποιητικά ανά την Ευρώπη. όπως ορίζεται με τα MOOS, τα Massive Online Open Courses ε, και άτυπες μορφές ε, μάθησης ώστε να μπορούν οι νέοι να συμβάλλουν σε όλο την Ευρώπη με τις γνώσεις και τις αξιότητες τους. Αυτές είναι κάποιες από τις κατευθύνσεις τις οποίες δεν θέλω να στην έκθεση. Εν γέννη θεωρώ ότι είναι καλή η έκθεση και αποτελεί ε, και χρειάζεται μόνο κάποιες ε, μικρές διευθετήσεις και μικροδιορθώσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πάβελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κρασνιτέτσκι τον εισηγητή για την καλή του έκθεση, ιδιαίτερος για την ε, δεκτική προς όλους προσέγγιση κατά την επεξεργασία των προτάσεων. Πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδιαίτερα δε για τη δημιουργία υψηλής ε, ποιότητα θέσεων εργασία. Η υποστήριξη που διατίθεται όμω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν έχει την ίδια, τα ίδια επίπεδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω γραφειοκρατικών διαφορών και, απουσία, και λόγω απουσίας ε, ασφάλειας δικαίου και σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία τη σχετική με την ιατροφαρμακευτική περιθάλψη και την συνταξιδοτική ασφάλιση. Στι τροπολογίε μα θα ζητήσουμε ισότιμη πρόσβαση στην ε, μικροχρηματοδότηση και τι πιστώσει, υποστήριξη για τι νεοφυεί επιχειρήσει, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό τους για δημιουργία νέων θέσεων Θέλουμε να αναπτυχθεί επίσης από τα κράτη-μέλη ενεργός πολιτική για την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και οι υποδομές εκείνες που θα ενθαρρύνουν και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω πως ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν εταιρικές σχέσεις, επιχειρηματικές σχέσεις, συνδικάτα ε, οργανώσει των πολιτών και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της ποιότητας των ε, προγραμμάτων δράσεως. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για την ε, μεταλλαγή του συστήματος ε, εργασίας στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κανονιστικό σύστημα για τις κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάπαλοβα, τρίτη σκιώδης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση και την επισκόπηση. Συμφωνούμε με τα προστασία του σχεδίου. Η κυρία Χάρκινο, συντονίστρια, έχει την ε, ευκαιρία να περιγράψει τις κυρίες θέσεις της Άλντε και τις δικές μου βέβαια, όταν εγώ δεν ήμουν παρούσα. Δυστυχώς χρειάστηκε να αναβληθεί αυτή η δουλειά, δεν μπορούσα όμως να κάνουμε τίποτε διαφορετικό. Και το μεταξύ έχω καταθέσει μας με τους συναδέλφους τροπολογίες, θα σας ενημερώσω μόνο ε, για ορισμένες από αυτές, όπου ζητούμε επί παραδείγματι προαγωγή της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, όπως είδατε και χτες ε, στην μεικτή μας συνεδρία με την Επιτροπή Πολιτισμού. Με χαρά διεπιστώσαμε πως και οι δύο επίτροποι έχουν καταστήσει τη διάσταση αυτή προτεραιότητα και μέσα στο νέο θεματολόγιο δεξιότητων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Επίση σταθερό αλλά και ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον είναι απαραίτητο, όπως πολύ σωστά ε, ε, επισημαίνει και ο ε, εισηγητής χρειάζεται ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον για να μπορούν να λειτουργούν και να συνεχίζουν να αναπτύσσονται οι καλύτεροι, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη για τις νεοφυείς, τις μικρομεσαίες, τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες θα μπορέσουν να αναπτύξουν τι δραστηριότητε του και να απασχολήσουν υψηλή ε, δεξιότητα δυναμικό. Οι μικρομεσαίε θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μείωση του κόστου χάρη στην ψηφιοποίηση και κυρίω ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, το ηλεκτρονικό σύστημα η e-government δηλαδή, για να μπορέσουν να απτύξουν το μέγιστο την ε, το δυναμικό για την ανάπτυξη της συνεργασίας. Και βέβαια θα σα ξαφνιάσει το γεγονό ότι πρόκειται να καταθέσω ε, τροπολογίες για τα συστήματα μαθητείας ε, ασκουμένων και ούτω καθεξής που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία λοιπόν και προσβλέπω στην ε, συζήτηση του τελικού, της τελικής εκδοχής της έκθεσης. Η Πρόεδρος, ο κύριος Ηλικιώτης δεν είναι εδώ, θα τον εκπροσωπήσετε εσείς, μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαβάσω την δήλωση του κυρίου Σιλικιώτη για την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εμπλοκή του και την συνεισφορά του. Και φυσικά η πολιτική μας ομάδα σκοπεύει να συνεργαστεί μαζί του με στενό τρόπο. Συμφωνούμε με την αντίληψη ότι οι μικρομεσαίες θα πρέπει να προστατευτούν καλύτερα διότι αποτελούν τον σκελετό της οικονομίας. Αλλά οι σκιώδεις της ΓΚΟΕ δεν είναι βέβαιοι αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα τομέα μικρομεσαίων. Το θέμα επίσης του λεγόμενου κόστους της εργασίας ε, θεωρείται ένα βάρος για τις μικρομεσαίες, της παραγράφους 3 και 13. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Να μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες δεν θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κοινωνικό ντάμπινγκ το οποίο επιβάλλουν και προωθούν οι, μικρομεσαίες, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως σωστά λέτε στην παράγραφο 4. Υπάρχει, θα έλεγα, ένα ιδιαίτερο βάρος για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι τόσο στα συμφέροντα γενικότερα των μικρομεσαίων. Πάντως θα συζητήσουμε τις παραγράφους μία προς μία, θα καταφέσουμε τροπολογίες και θα συζητήσουμε και τις προτινόμενες συμβιβαστικές. Thank Σας ευχαριστώ. Ζντάνοκα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και μια πολύ καλή έκθεση σημαντική έκθεση για την προώθηση επίσης του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και την δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι πράγματι θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα συμφέροντα των εργοδοτών Ξέρουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος στις μικρομεσαίες δεν είναι και τόσο διαδεδομένος όσο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αναφερόμαστε σε διαφορετικές μορφές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα θέλαμε να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά, ειδική αναφορά και σε ε, Εταιρείε συνεστεριστικού χαρακτήρα, συνεργατικού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους και μέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σαν λογική όταν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μειώνουν τις αμοιβέ και όχι τον αριθμό των εργαζομένων. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση αυτή και θα συζητήσουμε στα σημεία που υπάρχει διαφωνία με τον εισηγητή. Thank ευχαριστώ. Η κυρία Ατζουά δεν είναι εδώ. Άρα το λόγο έχει ο Ντομινίκ Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα όχι μόνο να ευχαριστήσω τον κύριο Κρασνοντεύσκη, αλλά να τον συγχαρώ. Πραγματικά. Διότι το γεγονό ότι τοποθέτησε στο κέντρο του συστήματος τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 80 με 90% του μεγέθους, του πληθυσμού του συνολικού που ασχολείται στις επιχειρήσεις, το γεγονός ότι τις τοποθετεί λοιπόν στο κέντρο του συστήματος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, είναι στην καρδιά του προβλήματος και αντιπαρατίθεται με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις να αποφύγουν κάθε άκτος, κάθε φορολογική επιβάρυνση, κάθε συνεισφορά. Οι τράπεζες, τα πιστοτικά ιδρύματα υποστηρίζουν άλλα πιστοτικά ιδρύματα και καμιά φορά τις πολυεθνικές. Περνώντας από τις επενδύσεις τις εθνικές και τις περιφερειακές. Τίποτα για τις ΜΜΕ. Και οι καθυστερήσεις πληρωμών που καθυστερούν 60, 70, 80, 90 μέρες γιατί πολύ συχνά ξέρετε στην αλυσίδα της υπεργολαβίας συμμετέχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η συνεισφορά τους στην τελική, στον τελικό καθορισμό της τιμής που τελικά επιβαρύνει τον καταναλωτή, η συνεισφορά τους είναι πάρα πολύ μικρή. Όμως, φοβούμε ότι πάλι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κάπως αντίστροφα. Δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λέτε για να δημιουργήσουν εκείνες θέσεις απασχόλησης. Το πραγματικό ερώτημα θα ήταν πώς να τις βοηθήσουμε να μην καταστρέψουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης. Γιατί αν πάρουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα της Γαλλίας, χίλιες θέσεις την ημέρα χάνουμε από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τους μικρούς βιοτέχνες, από τα συνεργεία αυτοκινήτων, από τέτοιου είδους μικρές επιχειρήσεις. Ανακοινώνουμε στα νέα και στις ειδήσει για τις περικοπές που κάνουν μεγάλη όμιλη, αλλά δεν διαβάζουμε για τη σώρευση όλων αυτών των θέσεων απασχόλησης που χάνουμε από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, το κέντρο βάρους μας θα, ήταν, θα έπρεπε να είναι περισσότερο ως αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κρασνοντέψκι θα ήθελε να πει δύο λόγια. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ναι, με συγχωρείτε, έχω λησμονήσει δύο. Ο Τόμας Μάν είναι πρώτος. Πρόεδρε, ναι, ζητήσαμε το λόγο. Γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο κύριος Κρασοντεύσκη το γνωρίζει πολύ καλά. Και μια και γνωρίζει και τη γλώσσα μου, όταν έχουμε την ευκαιρία στο αεροπλάνο να συναντηθούμε, ερχόμενοι στις Βρυξέλλες, συζητούμε συχνά τα θέματα. Αυτά είναι πολύ καλή έκθεση, λοιπόν. Το είπα και στους συναδέλφους από την ομάδα μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να μην λέμε μόνο πόσο δύσκολο είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά πάνω απ' όλα τι είδους δυναμικό διαθέτουν αυτές και το έχει περιγράψει εξαιρετικά. Το brain drain, η διαρροή εγκεφάλων, ένα τεράστιο θέμα και το έχουμε πολλές φορές επισημάνει. Ε, θέλουμε να φτιάχνουμε επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση με τον εργαζόμενο, τον εκπαιδεύουν πολλές φορές, αλλά μετά τι γίνεται. Όταν κάποιος ε, δηλαδή μπορεί να αναζητήσει διαφορετικά ε, την τύχη του. Και επίσης πολύ συχνά υπάρχει η παράλληλη οικονομία, η σκιώδης οικονομία. Δρά και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει ή δεν θέλει να την ελέγξει. Εμείς πιστεύουμε στην αξία και τη δύναμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να δρουν μέσα σε ένα ε, θεμητό πλαίσιο. Και όταν μιλούμε για μικρές και μεσές επιχειρήσεις, έχουμε επιχειρηματίες μικρομεσαίους που στο παρελθόν είχαν Τριετέ και πενταετέ ακόμη πρόγραμμα για τις εταιρείε τους. Τώρα πια αυτό δεν είναι δυνατόν και καλούνται να γίνουν ευέλικτοι όπως και εμείς σε κάθε τομέα, ακόμα και στους πόρους, γιατί αυτό η, η, η σταθερότητα πια δεν υπάρχει. Ζητήματα κατάρτισης, εκπαίδευσης, ε, απόκτησης δεξιοτήτων έχουν πολύ μεγάλη σημασία ώστε να μπορούμε και εμείς ε, να βοηθούμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προφροντίζουμε εμείς από τον κοινωνικό τομέα να ε, διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νέους. Βλέπω στη χώρα μου ενώσεις για την απασχόληση με προσπάθειες για την εξασφάλιση συμφώνων ε, για την κατάρτιση. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε ίσως να δώσει αποτελέσματα και σε άλλες χώρες. Μια συμμαχία δηλαδή για τους νέους που θα τους προσφέρει μια πραγματική και ουσιαστική ευκαιρία και ολοκληρώνω πρόεδρε. Η κοινωνική ευθύνη δεν θα πρέπει να είναι για τις επιχειρήσεις ένα άλοθη, αλλά μια προγραμματική, μια σημαντική θέση, δηλαδή με αυτή να λένε ότι θέλουν να επιτύχουν περισσότερα. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απλώ ιδεαλιστές και εγώ δεν είμαι ρομαντικός. Έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ε, πειραματικά ε, εγχειρήματα και που έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θετικά. Θα προσπαθήσω με κάθε δύναμη να υποστηρίξω και ε, την έκθεση σας και περιμένω 12 η ώρα της 27 Απριλίου πώς και πώς. Thank you. I... Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σόντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για την γνωμοδότηση αυτή και για το θέμα αυτό που μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Ε, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή ε, για την δουλειά του αυτή που μας βρίσκει σε πάρα πολλά σημεία σύμφωνους και εγώ συμφωνώ για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ε, απασχόλησης, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον πολύ σημαντικό ρόλο, τον εδαφικό και τοπικό και περιφερειακό ρόλο που έχουν στην μετάδοση της γνώσης, στη μετάδοση της τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα προγράμματα κατάρτισης και ασκήσεως. Δύο λοιπόν στοιχεία που αναφέρει η έκθεση είναι καταρχάς οι αξίες της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν που θα πρέπει να περνούν από τα εκπαιδευτικά συστήματα και από τα συστήματα κατάρτισης ώστε όλα αυτά να μην μένουν στα λόγια αλλά να γίνονται πράξη να γίνονται δραστηριότητα επιχειρηματική και δημιουργία αλλά θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το ρόλο που έχουμε εμείς εδώ να διαδραματίσουμε, το ρόλο δηλαδή που έχει να διαδραματίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, πρέπει να είναι αυτό σταθερό, αυτό υπόθηκε, και θα πρέπει να σταματήσουν τα κράτη-μέλη να υπερνομοθετούν, να υπερρυθμίζουν, γιατί αυτά είναι εμπόδια και περιορισμοί για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης αυτές οι επιχειρήσεις να λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία του σχεδιασμού της πρότασης νέας νομοθεσίας από την πρώτη στιγμή που σχεδιάζουμε τις νέες νομοθετικές προτάσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την νομοθεσία στην περίπτωση των ΜΜΕ. Αυτό ακόμα πιο συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των τριμερών διαλόγων μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασναντεύσκη έχει ένα σύντομο σχόλιο από ό,τι κατάλαβα. Πρωτού συνεχίσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και για τις επικρίσεις τους και για τα επικοδομητικά τους σχόλια και για τις προτάσεις και ιδέες τους. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία και ένα συμβαστικό, μια συμβαστική πρόταση κειμένου. Εγώ στα πλαίσια της μελέτης αυτής μίλησα με μικρούς παραγωγούς, με μικρούς βιοτέχνες, από όλους τους κλάδους μου διηγήθηκαν τα προβλήματά τους, μου εξήγησαν ποια είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Και όπως ε, λέει και ο κύριος Μαν, ανεξαρτήτως του ποια είναι η πολιτική ομάδα και η ιδεολογική τοποθέτησή μας, μπορούμε να βρίσκουμε κοινό τόπο. γιατί έχουμε την ευκαιρία να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, να καταλάβουμε καλύτερα τις διαδρομές που έχουμε διανύσει. Να μιλούμε περισσότερο για τις εμπειρίες των χωρών μας. προκειμένου να δημιουργούμε την Ευρώπη από κοινού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρασναντεύσκη. Η συζήτηση αυτή θα ακολουθηθεί τώρα από μια παρουσίαση για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις μικρομεσαίες. θα έχουμε αν θέλετε ε, το θέμα τώρα ειδωμένο από διαφορετική σκοπιά, όχι από πολιτική σκοπιά, αλλά από πιο τεχνική. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάντελ, στην κυρία Μάντελ, υπεύθυνη για το Eurofound για την αναζήτηση εργασίας. Δημιουργία λοιπόν θέσεων απασχόλησης για τις μικρομεσαίες. Έχετε το λόγο κύριε Μάντελ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την έρευνα αυτή. Είναι ένα θέμα σημαντικό νομίζω για όλους που έχει ήδη συζητηθεί και θα συνεχιστεί η συζήτηση γι' αυτό. Όπως επανειλημμένα έχει υποθεί, οι μικρομεσές δεν είναι μόνο σκελετός της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά θα συνεισφέρουν σημαντικά στον δυναμισμό της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat το 2014, είδαμε ότι για πρώτη φορά μετά από την αρχή της χρηματοοικονομικής κρίσης άρχισαν οι μικρομεσές να προσλαμβάνουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι υπεύθυνε και για τη μεγάλη πλειοψηφία των θέσεων απασχόλησης το 2014 και υπάρχουν καλές προβλέψεις και για τον προηγούμενο χρόνο. Είναι μια θετική λοιπόν πλευρά, να μην μιλάμε μόνο για τα προβλήματα των μικρομεσαίων αλλά και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στις ε, μικρομεσαίες μεταξύ τους. Δεν αναπτύσσονται όλες οι μικρομεσαίες, αν και όλες θέλουν να αναπτυχθούν. Έχουν ε, πάντως ικανοποιητικές επιδόσεις και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μεταξύ τους διαφορές. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Να δούμε ποιες είναι οι μικρομεσαίες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να ανταπτυχθούν και σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθηθούν από το ε, κρατικό ή το κοινοτικό πλαίσιο. Ανάμεσα στη μεγάλη λοιπόν ποικιλία των μικρομεσαίων, ποιες είναι οι πιο δυναμικές σε σχέση με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και αν κάποιες το πετυχαίνουν αυτό, γιατί κάποιες άλλες αποτυγχάνουν στην ίδια προσπάθεια. Όλα αυτά τα θέματα μπορεί να οδηγήσουν στην βελτίωση των πλαισίων στήριξης ε, για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν έχει συζητηθεί επί μακρόν ποια είναι τα εμπόδια και τι λειτουργεί σαν τροχοπέδι στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έχουν γίνει κάποιες επιμέρους συζητήσεις, ειδικά για τους διαφθρωτικούς δείκτες. δείκτες ε, χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη είναι όπως η ηλικία της επιχείρησης, οι νεοπαγείς επιχειρήσεις, οι νεοφυείς επιχειρήσεις ε, δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, είναι λογικό. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Οι παλιές δεν δημιουργούν και οι καινούργιες δημιουργούν, είναι πολύ πιο περίπλοκα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια τα οποία επηρεάζουν και εδώ οι δείκτες είναι περίπλοκοι. Κάποιοι δείκτες εδώ είναι εκτός της επιχείρησης, το μπλε τμήμα του πίνακα και από την άλλη είναι οι δείκτες οι οποίες επηρεάζονται και επηρεάζουν με τη σειρά τους την οικονομική ανάπτυξη των, μικιών, των μικρομεσαίων. Θέματα όπως η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, τα διοικητικά βάρη κτλ. Βέβαια αυτοί οι παράγοντες είναι ένα μόνο κομμάτι της ιστορίας, υπάρχουν και πιο σημαντικά θέματα όπως ο ρόλος του εργοδότη, του υπεύθυνου της επιχείρησης, οι δεξιότητες τις οποίες ε, έχει, η καινοτομική διάθεση, η δυνατότητα να διατρέξει κινδύνους για να πετύχει τους στόχους, Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι μεταξύ τους επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και ενδιαφέρουν από τη μία επιχείρηση στην άλλη. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν είναι να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων στην Ευρώπη. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε εδώ απλή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι νέε αναπτύσσονται και οι παλαιέ όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, είναι πολύ παραγοντικό το σύστημα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το προφίλ μιας τέτοιας καταρχάς επιχείρησης. Προσπαθούμε να δούμε ε, ποια είναι η επιχείρηση η οποία δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες όπως βλέπετε που επηρεάζουν την δημιουργία ηλικία, εθνικοί παράγοντες, διεθνείς παράγοντες, δευτερεύοντες παράγοντες. Πρέπει να υπάρχει επιθυμία να διατρέξουν κάποιο οικονομικό κίνδυνο, πρέπει να υπάρχει η επιθυμία βελτίωσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και η δυνατότητα σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μια επιχείρηση ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει την εικόνα της ελκυστικής επιχείρησης στην αγορά εργασίας για να μπορεί να προσελκύει πρόσωπα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και να ανταγωνίζεται έτσι τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είναι κατά συνθήκη πιο ελκυστικές. Όπως βλέπετε όλα αυτά είναι περίπλοκα και όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα για την επιχείρηση και για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον τρόπο συνεπώς στήριξή τους. Το θέμα δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και θέμα ποιοτικό των θέσεων απασχόλησης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στις μικρομεσαίες αυτές. Βλέπουμε και εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές βλέπουμε εδώ μια διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Βλέπετε ε, στις γκρίζες στήλες τις θέσεις ε, εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης και από την άλλη τις θέσεις απασχόλησης ε, που δημιουργούνται μετά. Στις μικροεπιχειρήσεις βλέπουμε να υπάρχει μια συνολική μείωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ενώ στις μικρές επιχειρήσεις ήδη διαφαίνονται κάποια δείγματα δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. και σε επίπεδο χαμηλά αμοιβωμένων θέσεων και σε επίπεδο υψηλά αμοιβωμένων στελεχών δηλαδή ε, των εταιριών αυτών. Έχει σημασία επίσης γύρω από το θέμα αυτό να δούμε ότι η έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη. Επιμέρους και διάσπαρτα είναι τα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή μας και γι' αυτό και τα ευρήματά μας είναι και αυτά περιορισμένα και πολυδιασπασμένα. Βλέπουμε ότι σε κάποιους τομείς οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν καλύτερα από τις μεγάλες, σε κάποιους άλλους τομείς όχι και οι δύο μπορούν να έχουν δίκιο γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε επίσης ανάγκη από περισσότερους σταθερούς δείκτες όπως οι αμοιβέ, η αντιπροσωπευτικότητα. Φαίνεται ότι ε, εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η αξιολόγηση, το υποκειμενικό της ε, θέσης εργασίας, της εκτίμησης της εικόνας φαίνεται ότι είναι υψηλότερο και καλύτερο στις μικρές από ό,τι στις μεγάλες. Ένα άλλο θέμα που θέλησα να ερευνήσω είναι το ποια είναι η διαδικασία για την δημιουργία της θέσης απασχόλησης. Το πρώτο έβριμα εδώ και δεν εκπλήσει είναι ότι ε, αυτό γίνεται ανεπίσημα στις μικρομεσαίες. Ε, στην ουσία γίνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία δημιουργίας θέσης απασχόλησης. Σε σχέση βέβαια με άλλες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στις μικρομεσαίες, το θέμα αυτό αποτελεί στρατηγικό παράγοντα. θέλουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι βιώσιμες, να είναι μακροπρόθεσμες και ε, να μπορέσουν σαν επιχείρηση να έχουν την δυνατότητα μακροπρόθεσμης κάλυψης της δαπάνης αυτής. Τώρα αναφερθήκατε σε κάποια άλλη φάση των συζητήσεών σας σε ατυπικές μορφές γνώσης και ικανοτήτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην διαδικασία προσλήψεων στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις ε, ε, τα curriculum vitae και τα διπλώματα έχουν μια κάποια σημασία, αλλά φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι οι συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις είναι το βασικό στοιχείο και χαρακτηριστικό και ακριβώς πολλές φορές δεν αρκεί μία συνέντευξη, αλλά χρειάζεται μία ολόκληρη σειρά συνεντεύξεων, τέσσερις ή πέντε, δεν εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία αυτή μόνο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή μόνο ο μάνατζερ του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, αλλά πολύ μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων. Αυτό το οποίο βιώνουν λοιπόν είναι μία αμφισβήτηση της διαδικασίας πρόσληψης. Αν δεν βρίσκουν τις, ε, τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουν στην αγορά εργασίας, τότε προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο κατάλογο απαιτήσεων πιο διαρθρωμένο στη δεύτερη φάση. έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα και το μισθολογικό κόστος. Για να τελειώσω, εδώ βλέπουμε κάποιους δείκτες που είναι χρήσιμοι για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, φυσικά είναι το γραφειοκρατικό βάρος, το οικονομικό κλίμα, το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν επίσης και κάποια επιμέρους δευτερεύοντα στοιχεία όπως ακριβώς αυτό το οποίο είπα, το επιχειρηματικό πνεύμα, η κουλτούρα του να διατρέξει κανείς, να αναλάβει να διατρέξει κάποιον οικονομικό κίνδυνο για να πετύχει. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενα αρρωγής προς τις μικρομεσαίες, όχι υποχρεωτικά από τις κρατικές υπηρεσίες. Πολλές φορές οι οργανώσεις των μικρομεσαίων είναι ισχυρές σε διάφορες χώρες και βοηθούν τις εταιρείες, διότι κατέχουν την τεχνογνωσία για να το κάνουν. Σε κάποιες από τις χώρες αυτές το κλίμα για την ανάπτυξή τους όμως δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό και ε, η σημασία εδώ είναι ακριβώς να βελτιωθεί ο τρόπος στήριξής τους. Τα θέματα της αγοράς εργασίας είναι σημαντικά και συνδέονται με τις προσλήψεις, επίπεδο μισθών, γκρίζα οικονομία, ανταγωνισμός μεταξύ τους των μικρομεσαίων, εργατική νομοθεσία, η οποία μπορεί να είναι ειδική για τις μικρομεσαίες ή γενικότερα να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και οι δεξιότητες οι οποίες πολλές φορές δεν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τις οποίες έχουν οι μικρομεσαίες και εδώ τίθεται σε αμφισβήτηση ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος κατάρτισης. Από την άλλη οι μικρομεσαίες είναι καλές για να κάνουν εκπαίδευση των εργαζομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης και να προσλαμβάνουν και μαθητευόμενους που θα στηρίξουν καλύτερα τις ανάγκες τους και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και τώρα, για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Είδαμε όλα αυτά τα στοιχεία, είδαμε πώς επηρεάζουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, είδαμε όλα τα επιμέρους και διαφοροποιούμενα μεταξύ τους χαρακτηριστικά και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια μονοδιάστατη μορφή στήριξης, ένα μονοδιάστατο μέσο στήριξης. Νομίζω ότι εδώ τίθενται πολλά πρακτικά θέματα, όπως και το θέμα του one-stop shop. Ίσως θα πρέπει να σταματήσω εδώ σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγή έμπνευση στα όσα μας είπατε. Δεν φαντάζομαι να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Ωστόσο, αν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να διανύμουμε την εκθεσή σας στα μέλη της Επιτροπής, μια και αρκετοί έχουν ήδη αποχωρήσει. Θα είναι χρήσιμη, πιστεύω. Σας ευχαριστώ θέρμα για την παρουσία εδώ και την παρουσίαση. Ε, I just also want to remind you that, ε, Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι 27 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. 30 Μαΐου εξετάζω την τροπολογία στην έκθεση Κρασνιεύσκη. 15-16 Ιουνίου η έγκριση στην Επιτροπή και συζήτηση στην Ολομέλεια του Σεπτέμβριου. Και έτσι περνώ στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την κοινωνική ενσωμάτωξη και έντοξη στην αγορά εργασίας εν ώψη της εκθέσεως πρωτοβουλίας για τους πρόσφυγες. Ξεκινώ. Δίνοντας το λόγο στην κυρία Μανουέλα Γκελένα της Επιτροπής. Και βεβαίως ο συντάκτης και οι σκιώδεις μπορούν να λάβουν το λόγο. Ξεκινώ όμως με την κυρία Γκελένα παρακαλώ. Πρόεδρε, η κυρία Γκελέγκ δεν είναι παρούσα. Έγινε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμά τη και έτσι την αντικαθιστώ εγώ. Α, πολύ ωραία λέει η πρόεδρο. Παρακαλώ, όπω και να σα λένε, πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ. Ξεκινώ με ορισμένε σκέψει για το ζήτημα ενσωμάτωση στην αγορά εργασία ε, προσφύγων και ετούν άσυλο Εκπροσωπώ βεβαίω τη Μανουέλα και την Task Force ομάδα κρούσεως για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασία που θεσπίστηκε σε επίπεδο Επιτροπή και, και δει στην Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, DG Employment. Η ενσωμάτωση στην αγορά εργασία είναι βέβαια αρμοδιότητα κατά κύριο και πρώτο λόγο των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει να προσφέρει υποστήριξη και κίνητρα στι δράσει των κρατών μελών, επί παραδείγματι προάγοντα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρώιμη ενσωμάτωση στην αγορά εργασία και ε, κοινοτική χρηματοδότηση. Η κατάσταση των προσφύγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απαιτεί περισσότερες φιλοδοξίες και συντονισμένες δράσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής και ιδιαίτερα την απασχόληση, την εκπαίδευση, κοινωνική συμπερίληψη, ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων. Ε, πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν καθώς και από την ανταλλαγή των πρακτικών και εμπειριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πέραν τη κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, απαραίτητο είναι προαχθεί η ενεργό συμμετοχή του στη χώρα υποδοχής και κυρίως η ένταξη τους στην αγορά εργασία. Η αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασία έχει ρόλο κλειδί και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, ναι, για να εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό να εξασφαλίσουν ότι οι αιτούντε άσυλο θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία εντό εννέα μήνου από την υποβολή αιτήματο διεθνού προστασία. Ορισμένα κράτη-μέλη επιτρέπουν στου αιτούντε το άσυλο να ενταχθούν στην αγορά εργασία ακόμη νωρίτερα φέρει πίν η Σουηδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία δίνουν άμεση πρόσβαση. Η Αυστρία και η Γερμανία μέσα στο τρίμηνο, το Βέλγιο ύστερα από τέσσερι μήνε από την υποβολή τη έτσι για, διεθνή προστασία. Άλλοι ακολουθούν τα καλά παραδείγματα αυτά, όπω η Ιταλία που έχει περιορίσει από έξι σε δύο μήνε την περίοδο αναμονή. Για να διευκολυνθεί η ένταξη στην αγορά εργασία είναι σημαντικό να, εξασφαλιστεί, ε, να εξασφαλιστούν μαθήματα γλωσσών, εκπαίδευση κυρίως για τα παιδιά, κατάρτιση και βεβαίως θα πρέπει να επιταχυνθεί και η αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασία για τους πρόσφυγες και τούντε άσυλο, η α, α, ε, εκπαίδευση σχετική, η κατάρτιση σχετική με τις πολιτιστικές αξίες επίση χώρας υποδοχής έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να προαχθεί. Η ανταλλαγή λοιπόν ιδεών και βέλτιστων πρακτικών έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει επίση να επαναληφθεί η δέσμευση για την ένωση των δυνάμεων όλων των κρατών προκειμένου να ε, αποδεχθούν και να ενσωματώσουν στην αγορά εργασία του του πρόσφυγε και του δεσάσυλο. Πρόκειται για υπηρεσίε με πολύ μεγάλη σημασία ώστε να υπάρξει αυτή η αντιστοίχηση μεταξύ των ανέργων ε, και τη αγορά εργασία, ώστε να είναι γνωστέ οι ανάγκε τη αγορά εργασία και των ανέργων. Έχουν πολλέ δεξιότητε οι πρόσφυγε, μπορούν να συμβάλλουν στι οικονομίε των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι δεξιότητες απορροφώνται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα, υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση, γλωσσικές, ε, γλωσσική μάθηση παραδείγματι και ταυτόχρονα αναγνώριση και αξιού των δεξιότητων που ήδη διαθέτουν οι πρόσφυγες. Και όπως είπε χθε η Επίτροπος Τάισεν, η Επιτροπή σύντομα θα καταθέσει και θεματολόγιο δεξιοτήτων που θα περιλαμβάνει κεφάλαιο για τους πρόσφυγες. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να υποστηρίξει στη διευκόλυνση της εισαγωγής των μέτρων αυτών για ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νεοαφικθέντες αυτούς και αυτό μπορεί να το υποστηρίξουν και καθοδήγηση προς την πολιτική με βάση τις ε, ε, συστάσει ανακράτως μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. Επίση, ε, οι συνθήκε υποδοχή, αποδοχή ε, και ένταξη των ετούντων το άσυλο για το σημείο εισόδου, διελεύσεω ή τελικού προορισμού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι βέβαια όλοι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν έχουν επαρκή πόρου, γνώσει και ικανότητα γι' αυτό και έτσι συμβάλλουμε και εμεί με τα μέσα τα χρηματοδοτικά που έχουμε για να ενισχύσουμε τι δυνατότητε. Ε, αποδοχής και ένταξης των τοπικών αρχών στο προσωπικό το οποίο πρώτο υποδέχεται για να αντιμετωπίσει τις διάφορες πτυχές και τα περαιτέρω προβλήματα κοινωνικο-οικονομικά ως προς την ένταξη αυτών των υπηκών τρίτων κρατών και ειδικότερα των προσφύγων. Και τώρα θα περάσω σε αυτά τα οποία συγκεκριμένα πράττουμε εμείς στη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, μεταξύ των οποίων και τις δραστηριότητες της ομάδας κρούσεως Task Force. Αυτή η Task Force ασπίστηκε τον Οκτώβριο του 2015 Πέρσι δηλαδή. Ύστερα από ένα καυτό θα πω καλοκαίρι για την Ευρώπη σε σχέση με τα κύματα προσφύγων. Η βασική ιδέα ήταν να ε, Διόχετευθούν σε κατάλληλους διάβλους ήρωες ε, των μεταναστών και η απασχολησιμότητά τους σε διάφορους ε, τομείς και πέραν της Γενικής Διευθύνσης ε, για την απασχόληση και η συνεργασία μας βεβαίως με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις για το ίδιο θέμα αρμόδιες. Αυτό που κάνουμε εν προκειμένου είναι ότι συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση των Εσωτερικών Home αλλά και άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ιδιαίτερα δώσει έμφαση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμείνουν στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ε, προέλευση ε, και περιβάλλον μετανάστευση, αλλά και οι πρόσφυγες έχουμε για αυτό το λόγο αυτή την task force και όπως είπα και νωρίτερα κύρια ευθύνη για την ενσωμάτωση αγοράς εργασίας ανήκει στα κράτη-μέλη. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να συλλέξουμε και να προαγάγουμε ως το δυνατόν καλύτερες και πολλαποσχόμενες βέλτιστες πρακτικές για να τις διαθέσουμε διάγραμμικά σε όλους τους ενδιαφερομένους μπορούν έτσι να βρουν και να ακολουθήσουν τα καλύτερα παραδείγματα και αυτό είναι ένα εξελίξη έργο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε υποστηρίζοντα τα κράτη-μέλη στην ανταλλαγή των βέλτιστων και πολλά υποσχομένων πρακτικών και συγκεκριμένα ε, σκεφτόμαστε τη δυνατότητα εξασφάλισης ενός προγράμματος αμοιβαία εκμάθησης. Θα ξεκινήσουμε στις 22 Ιουνίου εδώ στις Βρυξέλλες με παρουσία της Επιτρόπου Τάισεν στην εκδήλωση που έχουμε σχεδιάσει και επίσης ε, διάφορα προγράμματα αμοιβαία μάθησης ή εκμάθησης που πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να υποφεληθούν με την ε, με το σύστημα των κοινών πρακτικών. Ιδιαίτερα η Ισπανία λοιπόν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και έτσι σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση το Μάιο. Υπάρχει επίσης ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας μέσα από το Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτούμενο για τους μετανάστες με όλες τις διαχειριστικές αρχές του Κοινωνικού Ταμείου, κοινωνικού εταίρους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες με στόχο την προαγωγή της αμοιβέ κατανόησης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρώτη συνάντηση το Φεβρουάριο εφέτος στις Βρυξέλλες. Όπως υπόθηκε νωρίτερα, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων τις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων, ιδιαίτερος δε όσον αφορά την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και προσπαθούμε να στηρίξουμε, να προσφέρουμε προστήριξη στις ε, ε, υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και για τον εντοπισμό και αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των προσφύγων και εν τέλει πολύ σημαντικό προσφέρουμε καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για την αξιοποίηση του ε, των κοινωτικών μέσων χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων. Για το συγκεκριμένο αυτό σημείο μπορώ να σα δώσω κάποιε περαιτέρω πληροφορίε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίε απασχόληση των ετούντων το άσυλο, όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήδη μπορεί να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη για την κοινωνική του ενσωμάτωση και ταχεία ένταξη στην αγορά εργασία τα μέτρα που προβλέπονται για την ένταξη των ε, ετούντων άσυλο και μεταναστών εν γέννη αφορούν ε, εκμάθηση γλώσσας, εντοπισμό αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση. Αυτά όμως μπορούν να χορηγηθούν μόνο στον ετούντα άσυλο που έχει νόμιμη και μόνο πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη ρητά χορηγούν στον ετούντα το άσυλο την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση ή σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των ανελίκων πέραν ε, της ατομικής υποστήριξης προς τον δάσυλο και την οικογένειά του μπορούν επίσης να ενισχυθούν οι διοικητικές δυνατότητες των υπηρεσιών των κρατών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται ιδιαίτερως με τις ειδικές ανάγκες και τις ε, ε, συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να αναζητήσουν μια διεθνή αναγνώριση για τις επαγγελματικέ τους ικανότητες, επίσης για τους, αυτού, αυτούς που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση. Ε, υπάρχει ένα μέτρο το οποίο επιτρέπει την υποστήριξη των ε, προσφύγων σε μια πρώτη υποστήριξη ε, με τρόφιμα, άμεση στέγη κτλ. Αλλά στην, σε επόμενο στάδιο αναγνώριση και νομικού καθεστώτου, στο βαθμό βέβαια που τα κράτη-μέλη έχουν εντοπίσει του ομάδε στόχου συγκεκριμένα και ζητούν την υποστήριξη του Ταμείου. Αλλά αυτά εξαρτώνται από το πεδίο που καλύπτουν τα εθνικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Πατρίσια Σιλβέρια και την Σουζάνε Γκράτς να μας δώσουν τις δικές τους ε, απόψεις, τη δική τους οπτική στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τη δουλειά μας ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης. Με δική μας ε, πρωτοβουλία έχουμε προετοιμάσει τρία keynotes για την ενσωμάτωση στην αγορά των ε, προσφύγων. Το πρώτο σημείωμα σχετικά με στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές έχει μία σύγκριση των προσεγγίσεων πολιτικής που έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί σχετικά με την κάλυψη ζητημάτων σημείων ε, που είναι ιδιαίτερως αμφίσιμα και προβληματικά. Το δεύτερο αναπτύχθηκε από έναν ε, σύμβουλο εμπειρογνώμονα ε, του οργανισμού σχετικά με την αποτελεσματικότητα του soft συντονισμού και το τρίτο αφορά στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκράτς που έχει προετοιμάσει τα κείμενα αυτά, τα σημειώματα αυτά για να σας μιλήσει για τα βασικά πορίσματα. Ευχαριστώ Πατρίσια. Αυτό που μπορώ να κάνω στα υπολοιπόμενα 8 λεπτά είναι μόνο να αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία για τις βέλτιστες ε, πρακτικές και την ενσωμάτωση στην αγορά των προσφύγων. Αυτό ε, το προετοίμασε το Ινστιτούτο απασχόλησης στη Γερμανία. Θα ήθελα να αφερθώ πρώτα σε κάποιες ποσοτικές πτυχές. Πρώτον, όλοι μιλούν για ένα κύμα προσφύγων. Αλλά τι σημαίνει αυτό για το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Ο ΩΣΑ μας δίνει κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι εάν ενσωματωθούν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο αυτό δεν θα είναι περισσότερο από το 0,4% του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Άλλο ένα μέγεθος προέρχεται από το Γερμανικό Ινστιτούτο, χώρα στην οποία είναι φιλότερος αριθμός των προσφύγων. Εάν λοιπόν υπολογίσει κανείς τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, έχουμε μια αύξηση του συνόλου του εργατικού δυναμικού κατά 1,5% σύμφωνα με τα μεγέθη του Ινστιτούτου. 1,5% λοιπόν πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Αλλά, και εδώ είναι άλλος ένας ε, παράγοντας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθότι η ενεργεία είναι, έχει κατέλθει, η επιρροή που μπορεί να έχει το μέγεθος των προσφύγων ή στη γερμανική αγορά και στη γερμανική ενεργεία μπορεί να είναι πιο σημαντική. Τώρα, έχουμε ενδείξεις ότι οι μετακινήσεις εντός της αγοράς εργασίας ε, μάλλον ε, μέχρι στιγμής ήταν ε, βραχή, διάρκεια, Μία ακόμα πτυχή σχετίζεται με το κόστος. Το κόστος για τα δημόσια οικονομικά μπορεί και να είναι σημαντικό έχουμε ενδείξει ότι θα μπορούσε να αφορά και στο 1% του προπολογισμού στην Σουηδία, 0,6% στη Δανία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σύμφωνα με τη μελέτη αυτές οι διακοιμάσεις έχουν και μία πτυχή ζήτησης και όχι μόνο προσφοράς. Η ενσωμάτωση δεν γίνεται δωρεάν πάντως. Ε, βλέπει κανείς τη μελέτη και το γνωρίζουμε και από άλλα διοικητικά στοιχεία στη Γερμανία, περί το 8% εκείνων που έχουν καταγραφεί με δημόσιες υπηρεσίες ε, κατάρτισης δεν έχουν πλήρη παιδεία, υπόβαθρο παιδείας ή κατάρτισης επαγγελματικής. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πρόσθετα κόστη κατάρτισης και χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα γλωσσικά μαθήματα. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων αυτών θα παραμείνουν για ένα παρατεταμένο διάστημα. Τι θα σήμαινε λοιπόν να μην τους ενσωματώσουμε, ποιο θα ήταν τότε το κόστος που θα έπρεπε να αναλάβουμε. Αυτά είναι τα ποσοτικά στοιχεία. Και θα σας δώσω ε, τους πέντε άξονες που καθορίσαμε μέσω εγγράφων πολιτικής από διάφορους φορείς και οργανισμούς. Καταρχά το έγγραφο που προετοιμάσει η DigiHome με τα εθνικά σημεία επαφής. Αυτό ήταν επί των μεταναστών, αλλά περιέχει και κάποια στοιχεία τους πρόσφυγες. Λάβαμε εγώ επίσης μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενσωμάτωση των προσφύγων η ο οργανισμός ε, United National Refugee και ένα έγγραφο του Διεθνούς Νομισμού Ταμείου. Δηλαδή, έχουμε μια κάλυψη και μια οπτική και ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών. Οι πέντε άξονες αυτοί είναι γνωστοί από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευρύτατη διεθνή συνένεση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, ακόμα και αν αυτό έχει κόστο. Καταρχά, η αγορά εργασία και η πρόσβαση. Οι νομικέ διατάξει και η υλοποίηση των οδηγιών ε, υποδοχή μπορεί να είναι εμπόδιο. Επίση, τα τεστ ή οι δοκιμέ απασχόληση, δηλαδή ότι οι πρόσφυγε μπορεί να προσληφθούν μόνο εφόσον δεν υπάρχει πολίτης της χώρας ή άλλος πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υποβάλλει ή περιορισμοί σχετικά με το ότι δεν μπορούν να είναι αυτοαποσχολούμενοι. Αυτά είναι περιορισμοί στην πρόσβαση και στην ταχεία ενσωμάτωση. Και γι' αυτό θα έπρεπε να έρθουν. Για τις ίδιες τις στρατηγικές ένταξης, και τώρα μιλώ για τους πέντε άξονες, συνοψίζω ως εξής. χρειάζεται μια γλωσσική στήριξη, χρειάζεται μια παροχή συμβουλών ε, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για τον κάθε από τους ε, πρόσφυγες. Χρειάζεται αναγνώριση των ε, προσόντων ή των τίτλων ή των δεξιοτήτων που έχουν το από το εξωτερικό, αλλά αυτό εξαρτάται απολύτως από τη χώρα. Είναι πιο εύκολο με το σύστημα εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, ε, είναι πολύ πιο δύσκολο σε ένα πολύ ε, πιο αυστηρά ρυθμισμένο σύστημα όπως το γερμανικό. Χρειάζεται τρίτον βοήθεια στην αναζήτηση θέσης απασχόλησης και χρειάζονται και στοχευμένες ενισχύσεις. Δηλαδή, πρέπει να αποζημιώνονται μόνο σχετικά με ε, αναγνωρισμένη ταυτοποιημένη παραγωγικότητα, κάλυψη συγκεκριμένων στόχων παραγωγικότητας. Τα στοχευμένα μέτρα για τους πρόσφυγες είναι απαραίτητα βεβαίω εφόσον δεν ομιλούν την γλώσσα τη χώρα υποδοχή. Γιατί τότε τέτοια μέτρα μπορούν να είναι και αντιπαραγωγία. Ο τέταρτο άξονα αφορά στην ενσωμάτωση στο πλαίσιο των δημοκρατικών αξιών και της κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο των οποίων είναι ε, σωστό και χρήσιμο να συμπεριλαμβάνονται και μη καπαόμικρον, ε, και κάποια προγράμματα εθελοντισμού ή αθλητικές δραστηριότητες και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες από τους πρόσφυγες ώστε να έρθουν σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών της χώρας υποδοχής. Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας είναι για τις ανάγκες της προσωπικές, της υγείας και ιδιαίτερα τις ανάγκες των γυναικών προσφύγων διότι έχουμε ενδείξει ότι αυτές ενσωματώνονται πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχουν θέματα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, δεν έχουν όλοι οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες ίση πρόσβαση και μεταχείριση από τις υπηρεσίες αυτής. Επίσης το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών δεν έχει διαπολιτιστική αν θέλετε κατάρτιση και δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο πρέπει να μεταχειρίζεται τους ανθρώπους αυτούς. Ένα άλλο σημείο που είναι αρκετά πιο αντιφατικό είναι το χρηματοδοτικό. Και αφορά στην ίση μεταχείριση στα επιδόματα, τα κοινωνικά επιδόματα και τους ελάχιστους μισθούς, το επίπεδο των επιδομάτων. έχουν επικρατήσει σε κάποιες περιπτώσεις ειδικέ προϋποθέσεις για τους πρόσφυγες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια και στην περαιτέρω παρεμπόδιση στην εσωμάτωση ή στην αγορά. Υπάρχει τώρα και, υπάρχει και το σύνολο προϋποθέσεων των επιδομάτων αυτών. και θα έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους πρόσφυγε εφόσον δεν συμμετέχουν στα μέτρα αυτά. Και ένα άλλο θέμα που έχει κινήσει συζητήσει στη Γερμανία είναι το θέμα και η συζήτηση για τον ελάχιστο μισθό, για τον κατώτατο μισθό. Είχαμε μιλήσει και με τους συναδέλφους του ILO σχετικά με τους κινδύνους ε, social dumping και άλλων αρνητικών επιπτώσεων στην αγορά εργασία. Ή, στη ή στη μελέτη καθορίσαμε κάποιε προκλήσει και διατυπώσαμε κάποιε συστάσει για το επίπεδο ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή τη στιγμή ε, μα λείπουν συγκρίσιμα δεδομένα σε σχέση με την ε, ένταξη και την ενσωμάτωση των μεταναστών. Για τους πρόσφυγες έχουμε πολλά κενά ακόμα στις πληροφορίες που έχουμε διάθεσή μας, το οποίο με οδηγεί στο δεύτερο σημείο που ήδη αναφέρθηκε, όλοι μιλούν για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά δεν έχουμε επαρκείς ενδείξεις, ούτε εδώ. Θα χρειαζόταν μια πολύ πιο συστηματική συλλογή στοιχείων σχετικά με το τι πραγματικά λειτουργεί καλώς στα κρατημέλη. Και το τρίτο σημείο, η συνεργασία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μου οδηγεί και στο δεύτερο σημείωμα για τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τις πλατφόρμες. Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία και, και μεγάλο αριθμό διαφόρων δικτύων, δίκτυα μετανάστευσης, υπό την δέλτα Home, άλλα δίκτυα υπό την δέλτα Employment, έχουμε το δίκτυο PES, Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες Μετανάστες και σε τοπικό επίπεδο υπό το γύρο της μια ομάδα και μια άλλη για την ε, ε, κοινωνική ένταξη των ε, μεταναστών. Γιατί τα θέματα αυτά είναι κοντινά το ένα προς το άλλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάπως περισσότερες πληροφορίες και πληρέστερη γνώση σχετικά με τα ιδιαίτερα θέματα και διαφορές με τους μετανάστες. Πάντως πολλά από τα στοιχεία, πολλή από τη γνώση που έχει συλλεχθεί έχει χρηματο... και έχει χρηματοδοτηθεί από την ε, Κομισιόν έχει σε κάποιο βαθμό απολεστεί στην παρία. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο δεύτερο σημείωμα και θα συνοψίσω πάρα πάρα πολύ σύντομα κάποια στοιχεία και από το τρίτο σημείωμα για τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είπε η Κομισιόν, integration that needs at least to Από ό,τι φαίνεται χρειάζονται 5 με 6 χρόνια προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένες ενδείξεις για τους πρόσφυγες αλλά θα πρόκειται για κονδύλια τα οποία κυρίως θα βρίσκονται υπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ακόμα και αν τα κράτη-μέλη ε, διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τους πόρους αυτούς και έχουν αναλευθεί κάποια μέτρα, παραμένουν κενά εδώ. Διότι ίσως τα κράτη-μέλη με πιο δύσκολη αγορά εργασίας να αντιμετωπίσουν δίλημα. Χώρες όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζουν έλλειψη πόρων και αν χρησιμοποιήσουν περισσότερα κονδύλια του ESF, ίσως οι δαπάνες τους για τους πρόσφυγες μπορεί να είναι εις βάρος άλλων δαπανών μακροπρόθεσμα ανέργων, γιατί ήδη δεν έχουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν διάφορες λύσεις Μία πρόταση που είχε υποβληθεί ήταν η χρησιμοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών μέσων, όπως κονδύλια τα οποία θα απευθύνονταν στις τοπικές κοινότητες, στους δήμους, οι οποίοι άμεσα διαχειρίζονται και ασχολούνται με τους ε, πρόσφυγες. Δεν υπάρχει όμως ε, συζήτηση πολιτικής από αυτού ακόμα. Στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής ε, Απασχόλησης του Κοινοβουλίου. Η προηγούμενη πρόταση επαναλήφθηκε να αυξηθούν τα κονδύλια για το ESF σε ένα 35% τη συμμετοχή επί του προπολογισμού, ώστε να. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αν μακρηγόρησα. Σα ευχαριστώ που δεν μου διακόψατε, που δεν μου πήρατε το μικρόφωνο είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Okay. Um, uh, we have a... Thank you both. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που θίξατε από πλευράς μας. κάντε σύντομες παρεμβάσεις και ερωτήσεις ε, ταυτόχρονα. Και στο τέλος θα δώσουμε την δυνατότητα στις δύο ομιλήτριες να δώσουν απαντήσεις. Αλλά ένα-ενάμιση λεπτό. Μην παρουσιάσετε συνολικά τα θέματα και πραγματικά θέστε και τις ερωτήσεις σας γιατί αλλιώς δεν τα καταφέρουμε. In uh, two parts. Is that okay? Okay, then I'll give the floor first to the uh, rapporteur, uh, Mr. Benify. Ο κύριος Μποναφέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που οργανώσατε αυτή τη συζήτηση για το θέμα της κοινωνικής ένταξης και εργασιακής ένταξης των προσφύγων. Αυτό δείχνει τη μέγιστη σημασία που δίνουμε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Task Force για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Δεν είμαι ο μόνος εδώ που πιστεύει ότι είναι απαραίτητο εσείς από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης να υγείστε τις προσπάθειες και να έχετε ακριβώς και την οργανωτική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται. Όταν ε, εγώ είχα προχωρήσει στη σύνταξη της έκθεσής μου, χρησιμοποίησα τις εργασίες σας. Ευχαριστώ και τη συνεργασία σας και ιδιαίτερα τη συνεργασία της κυρίας Γκελέγκα που είναι απούσα. Νομίζω ότι η συζήτηση θα κρατήσει για αρκετό καιρό και για την επεξεργασία των προγραμμάτων και για την πολιτική επεξεργασία. Να ευχαριστήσω και για την παρουσίαση των δύο συγκεκριμένων εκθέσεων. Οι αναλύσεις και οι συστάσεις είναι πολύτιμες σε αυτές τις δύο συνθετικές αλλά εξαντλητικές ταυτόχρονα παρουσιάσεις. Το θέμα δεν είναι απλά το επίκαιρο του πράγματος, αλλά να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και την συμμετοχή των πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Να πω ότι έχουμε να κάνουμε ε, με δύο θέματα πάνω στα οποία έχει σταθεί και η δική μου έκθεση. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω τεχνική ανάλυση Είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε και στη δική μου έκθεση αρκετά στοιχεία από τις δικές σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας, σας ευχαριστώ και για την ταχύτητα με την οποία προχωρήσατε και καταστήσατε διαθέσιμες τις εργασίες σας. Για τα ευρωπαϊκά ταμεία καταρχάς Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα την ενισχύσουμε γι' αυτό. Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι είναι ανεπαρκείς, αυτό είναι σαφές, αν τα συγκρίνουμε με τα αιτήματα που υπάρχουν για διεθνή προστασία τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό έχει ήδη ε, γίνει αντικείμενο αναφοράς και η μετατροπή των προγραμμάτων αυτών πρωτοβουλίας σε ένα λεπτομερές και συνεκτικό σχήμα, σε μια στρατηγική δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει, η οποία είναι κυρίως προσπάθεια απλοποίησης για την πρόσβαση στα ταμεία και θα επιτρέψουμε στους τοπικούς εταίρους, της πόλης σαν παράδειγμα, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και κάποιους επιμέρους πόρους για την ένταξη των ετούντων ασυλό και προσφύγων. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας προσεκτικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει, έτσι ώστε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να φανούν ευαίσθητε και να μην μειώσουν τις διαθέσιμες προτάσεις, κάτι το οποίο θα είναι εις βάρος και των προσφύγων και των χωρών ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κύριος Μάνης Κιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημαντικό είναι ότι μπορούμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα και να καταστήσουμε σαφή τη βάση. Πάντοτε όταν μιλώ σε σχολεία, παραπέμπω σε έναν ξεσημείωτο λόγο, σε μια ομιλία σημαντική του Ζων Κέρ που μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης, όπου αναφέρθηκε σε αυτούς που δεν θέλανε πρόσφυγες που έχουν κάνει το αντίθετο από αυτό που έπρεπε, που κλείσανε σύνορα, τους είπε θυμηθείτε τι ήσασταν κάποτε, πώς ήσασταν εσείς που είχατε πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Το θέμα δεν είναι τι χρειαζόμαστε από το Σέγγεν, τι θέλουμε να διαφυλάξουμε, αλλά και το πώς με όλα τα κύρια οικονομικά προβλήματα θέλουμε να συμπεριφερόμαστε ένα στον άλλον. και ότι χρειάζονται στοιχεία πλέον μιας κοινή πολιτικής για το άσυλο. Αυτό χρειαζόμαστε και όχι μία πολιτική θριαμβολογίας και εγκατάλειψη του πλησίων. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Πονιφάη, έχουμε ήδη συζητήσει. Πολλές ιδέες μας είναι ταυτόσιμες. Και το πρώτο, και πρέπει και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο που είναι να να εργαστούμε, είναι βέβαια η εκμάθηση της γλώσσας. Όχι βέβαια με την έννοια της ε, τιμωρίας. Όχι θέλουμε να σας τιμωρήσουμε γιατί θα στη χώρα μας, θα συγκριτηθούμε. Αλλά σας βοηθάμε. Εμπλουτίσουμε τις γνώσεις σας και με αυτόν τον τρόπο σας καθιστούμε ικανούς να δράσετε αυτόνομα. Το να λέμε με δύο-τρία γλυκούλια θα τα βρούμε και θα συνοηθούμε δεν αρκεί. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτοί που έρχονται στη χώρα υποδοχής μπορεί να μην βρούνε, να μην μείνουν για αρκετό χρόνο. Οι διαδικασίες της αναγνώρισης κρατάνε πολύ καιρό. Εάν λοιπόν ξεκινήσουν μια κατάρτιση στη χώρα υποδοχής και μετά την εγκαταλείψουν για να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, πρέπει να έχουν μπορέσει να αποκτήσουν κάτι και την αναγνώριση βέβαια τη επιπλέον γνώση. Χαίρομαι που μιλήσαμε νωρίτερα για τι μικρομεσαίε, γιατί είναι αρκετέ μικρομεσαίε που λένε ότι ναι, μπορεί να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε του πάντε, αλλά τουλάχιστον να προσφέρουν μια δυνατότητα ε, μαθητείας. Και έτσι μέσα από αυτό να δούμε και τι δυνατότητες υπάρχουν, τι προσφέρεται, τι δυνατότητες έχουμε για ένταξη και κυρίω αναφέρομαι στου νεότερου από αυτούς, που είναι πολλοί. Πολλοί όταν προσφέρεται η μαθητεία λένε «Μα εγώ χρειάζομαι λεφτά, δεν μπορώ να το κάνω δωρεάν». Και αν του πούμε «Μα τι τα θες τα λεφτά» θα μου πούνε «Άμα πρέπει να ξεπληρώσω κάτι φίλου. Και αυτοί οι φίλοι είναι βέβαια οι λαθροδιακινητέ. Ε, σε αυτό θα μπορούμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουν και εκείνοι την προσπάθεια που θα καταβάλουν οι μικρομεσαίες από πλευράς τους. Και ότι μπορούν και αυτοί από πλευράς τους να συμβάλλουν, ανεξαρτό του κόστους. Είναι σημαντικό αυτό. Και εν τέλει θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βεβαίως μπορεί να συμβάλλει, το αναφέρατε κι εσείς, Είπατε, έγινε λόγος νωρίτερα όμως για την δημιουργία ενός επιπλέον ταμείου. Ναι, αλλά να μην αρχίσει αυτό να μοιράζει χρήματα δεξιά-αριστερά. Να είναι ένα ταμείο το οποίο θα στοχεύει σωστά πάνω στις ανάγκες. Είναι απολύτως απαραίτητο. Ιδάλλως, από το κοινωνικό ταμείο παίρνουμε ένα κομμάτι με ένα σαφή τίτλο για να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Και όπως είπα και νωρίτερα στην άλλη συζήτηση, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, δεν πρέπει να φέρουμε σε αντιπαράθεση τον άνεργο με τον πρόσφυγα που ψάχνει για δουλειά. Πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτές τις έννοιες και τις ευθύνες. Χρήματα πάντα θα υπάρχουν. Για τις καταστροφές θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα. Ναι, ναι, βλέπω, βλέπω. Είναι απαραίτητο να δείξουμε, και αυτό ελπίζω εγώ πραγματικά, ότι ποτέ δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τις ανθρωπιστικές μας αξίες. Ευχαριστώ, Στίβενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Έχω κάποια σχόλια και ερωσμένες ερωτήσεις. Ξέρω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια πρόκληση όλοι μας και ιδιαίτερα πρέπει να μιλήσουμε για επιλογές και στόχους. Τα κράτη-μέλη έχουν βεβαίως δυνατότητες και αρμοδιότητες. Τι ζητάμε όμως. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους και από όλα τα κράτη-μέλη. Για όλους δηλαδή πρόσφυγες και μετανάστες όταν μιλούμε για δικαιώματα και ευθύνε. πρέπει να συστήσουμε πώ θα προαχθεί η ενσωμάτωση, η ένταξη και αν αποτελεί δικαίωμα ή υποχρέωση προς τους πρόσφυγες. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλοδεχθούμε, να τους υποδεχθούμε και να τους προσφέρουμε όσο δυνατόν καλύτερε δυνατότητε ενσωμάτωσης στις κοινωνίες μας και στι αγορέ εργασία. Για να ενταχθεί όμω κανεί στην αγορά εργασία χρειάζεται δεξιότητε. Κάποιοι εκ των προσφύγων ήδη έχουν προσόντα και δεξιότητε. Αλλά χρειάζεται να εξετάσουμε περισσότερο εάν μπορούν να αξιοποιηθούν. Καταρχά, αν είναι σωστέ πληροφορίε. εάν μπορούν να επιβεβαιωθούν και αν δεν προσφέρονται κατάλληλες δεξιότητες, να προσφερθεί εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα στη γλώσσα, η εκμάθηση της γλώσσας. Όταν κανείς έρχεται σε μια περιοχή όπως η Φλάνδρα, Φερρυπίν του Βελγίου, πρέπει να μάθει τη γλώσσα, τα φλαμανδικά ή στη Βαλονία αντίστοιχα τα γαλλικά. Είναι καθήκον όσο και υποχρέωση του πρόσφυγα και του ετούντα το άσυλο να μάθει τη γλώσσα. Εμείς δεν τον υποχρεώνουμε να έρθει στις χώρες μας, δεν τον πιέζουμε αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις ευκαιρίες που του προσφέρονται εδώ, πρέπει να είναι και ε, διατεθειμένος να μάθει τη γλώσσα υποδοχής, της χώρας υποδοχής. Και άρα χρειάζεται να διαβάσει, να μελετήσει. Όπως είπα, για να μπορέσει να ενταχθεί ένας πρόσφυγας στην αγορά εργασίας, πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα, ένας Σύρος, ένας Ιρακινός, με δεξιότητες, ακόμη και διδακτορική διατροφή, ε, εάν δεν σε θέση να επικοινωνήσει στα Ολλανδικά, δεν θα μπορεί να εργαστεί. Φέρει πίνη σε ένα περιβάλλον νοσοκομιακό στη Φλάνδρα, θα έλεγα. Και άρα πρέπει να βρεθεί η αντιστοίχηση των αναγκών Δεν μπορεί ο καθένας από οποιαδήποτε χώρα και με οποιαδήποτε κατάρτιση να έχετε σε αναγνώριση ανεξέταστα των δεξιοτήτων. Χρειάζεται η αναγνώριση και των γλωσσικών αλλά και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Τώρα είναι καθήκον της χώρας υποδοχής να προσφέρει αυτή την επαγγελματική κατάρτιση θα γίνει όλη αυτή η δουλειά για την ενσωμάτωση από τη χώρα υποδοχής. Δεν θα πρέπει και ο πρόσφυγας να αποδέχεται τις βασικές αξίες της κοινωνίας υποδοχής, όπως ισότητα ανδρών και γυναικών και άλλες αξίες. Τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Χρειάζεται περισσότερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Χρειάζεται να δασκόμαστε από τις θετικές αλλά και, τα, και τις κακές εμπειρίες άλλων κρατών στο παρελθόν. Η ανταλλαγή αυτή των βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν είμαι βέβαιη. Και για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών θα ήταν καλό να δούμε πώς μπορεί η Ανατολή και η Δύση να συνεργαστούν, πώς θα εξεταστεί το ιδιαίτερο πρόβλημα των γυναικών προσφύγων. Γιατί ξέραμε ότι στο παρελθόν οι γυναίκες πρόσφυγες, οι μετανάστριες πείθονταν να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας για να διατηρήσουν τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας προέλευσης τους. Έτσι έμεναν στο σπίτι να μεγαλώνουν τα παιδιά και οι άντρες μόνο δούλευαν. Αυτό είναι λοιπόν ένα άλλο θέμα. Πώς θα ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, σας ευχαριστώ. Όχι πάνω από τρία λεπτά παρακαλώ για τις παρεμβάσεις σας γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουμε μιας και ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε. Χθες εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο και όταν βλέπω στις ειδήσει τον τρόπο με το θέμα αυτό παρουσιάστηκε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με το πώς αντιδρούσαμε γι' αυτό πριν δύο χρόνια. Είναι θλιβερή η πραγματικότητα και δεν θα συμμεριστώ δυστυχώς τον ενθουσιασμό κάποιων συναδέλφων γύρω από το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τους πρόσφυγες. Το ότι 0,4% του εργατικού δυναμικού θα περιλαμβάνει το 1 εκατομμύριο εργαζομένων δεν έχει καμία σημασία, γιατί αν ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τους πρόσφυγες έχει αλλάξει. Έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, ερωτήσεις μάλλον. Διαρωτώ με σε ποιο βαθμό θέλουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα, θέλουμε να γίνουν σε εθνικό επίπεδο ή μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο μπορεί να προτείνει ευρωπαϊκό. Υπάρχει το θέμα των δεξιοτήτων και της ανταπόκρισής τους στις τοπικές ε, ανάγκες, ε, γιατί είναι σαφές επίσης ότι είναι δύσκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα στα τυπικά προσόντα και δεξιότητες και τα ατυπικά. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτού του είδους υποστήριξη δεν είναι συνεχής και διαρωτώ με τι έχει γίνει, έχει κάτι αλλάξει. Ξέρουμε ότι οι πλατφόρμες αυτές είναι σημαντικό να είναι λειτουργικές και να βοηθούν τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Γκονσάλες Πένιας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία, για τις συστάσεις, για τα συμπεράσματα και οι προτάσεις αυτές θα βοηθήσουν, είμαι σίγουρη, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω ε, είναι το θέμα του υψηλού κόστους και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς στην ουσία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ε, ένταξη στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση αυτή είναι σωστή. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα δεδομένα που τις στηρίζουν, που τις τεκμηριώνουν έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτό το κύμα εναντίον των προσφύγων το οποίο φαίνεται ότι διαμορφώθηκε σε κάποιες από τις χώρες της Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε επίσης αν αυτό έχει σχέση και με τις περικοπές του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας σε διάφορες χώρες, σε χώρες όπως τη δική μου, την Ισπανία, όπου οι μετανάστες δεν παίρνουν ταυτότητες ε, κοινωνικής πρόνοιας και οι Ισπανοί όταν πηγαίνουν σε άλλες χώρες χάνουν την δική τους ταυτότητα ε, για ε, την πρόνοια, την κοινωνική κάλυψη και όλα αυτά επηρεάζουν και τα θέματα της δημόσιας υγείας και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν, ε, αν και είναι κορεσμένα τέτοιου είδους καταστάσεις. Και σε άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης ισχύει το ίδιο. Υπάρχουν παραδείγματα χρηστών πρακτικών σκανδιναβικών χωρών, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Γίνεται αναφορά και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση στην Πορτογαλία είναι χώρες οι οποίες ε, δέχονται αρκετούς πρόσφυγες, αλλά θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό έχει αναλυθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο των μεσογειακών χωρών, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις συστάσεις αυτές. Είναι ειδική περίπτωση της Ελλάδας, όπου ο αριθμός των προσφύγων στο ελληνικό έδαφος ε, προϊόν της συμφωνίας με την Τουρκία και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από τα μνημόνια απαιτούν συγκεκριμένες ε, προσαρμοσμένες για τις καταστάσεις ε, ε, προτάσεις. Αναφέρεστε επίσης τους κοινωνικούς εταίρους, γίνεται επίσης αναφορά γενικότερα στο θέμα της ένταξης των προσφύγων και υπογραμμίζεται ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Και στις προτάσεις του ΩΣΑ γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στους κοινωνικούς εταίρους και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν οργανώσεις όπως τα συνδικάτα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να ανταλλάξουμε και σε αυτό το επίπεδο τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε επίσης και σε θέματα όπως η οικογενειακή επανένωση ε, υπάρχουν, ε, να υπάρξουν ειδικά μέτρα για τις ε, φιλετικές διακρίσεις, τις διακρίσεις των φίλων μάλλον. Στην Ισπανία, σαν παράδειγμα, οι πρόσφυγες δεν συμμετέχουν, δεν περνούν όλοι από τα συστήματα υποδοχής και έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια δεύτερη φάση ενώ δεν έχουμε καθορίσει την πρώτη φάση, τη φάση της υποδοχής. Πάρα πολλοί χάνονται και ε, στην ουσία ε, πέφτουν θύματα ε, παράνομων πρακτικών αυτών οι οποίοι χρηματοδοτούνται για να τους πέρασουν. Κοιτάξτε, μιλάτε για πάνω από τέσσερα λεπτά. Ζητώ συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Έχει η Τζιν Λάμπερ το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις της ομιλήτριας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν διάφορα δικαιώματα που ήδη έχουν οι προσφυγές και οι τούντες άσυλο υπό την ευρωπαϊκή νομοθεσία και μάλιστα υπό την οδηγία για τα προσόντα για την οποία υπήρξα και η συγγήτρια στο πλαίσιο της συζήτησης ε, σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας. Ήθελα να αναφερθώ και για το ρόλο που διαδραματίζουν διαματίζει η διάρκεια παραμονής τους, η διάρκεια της άδειας παραμονής τους. Πώς αυτό επιδρά με την ε, συμπληρωματική προστασία που λαμβάνουν και πώς αυτό διαδρά με την πρόσβαση σε κατάρτιση, με την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ή πανεπιστημιακά προγράμματα. Με ικανοποίηση άκουσα την ε, αναφορά στα επίπεδα εισοδημάτων, γιατί γνωρίζουμε ότι σε, σε κάποια κράτη-μέλη αυτά τα εισοδηματικά επίπεδα είναι ανεπαρκή και για τους πολίτες τους ίδιους της χώρας. Αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ε, πού είναι το κέντρο βάρους μας στην καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα που απορρέουν και από κάποιες από τις προτάσεις Κομισιόν σχετικά με το κεκτημένο του ασύλου. Σχετικά με την ιδέα αυτού του καινούριου ταμείου, υπάρχουν κάποιες απορίες, πιστεύω. Γιατί έχουμε δει πώς νέα κονδύλια αποσπώνται από ήδη φυστάμενα ταμεία, χωρίς να έχουμε νέους πόρους. Και θα έπρεπε να δούμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι που να δίνει άμεση πρόσβαση στους δήμους και τις κοινότητες. Υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηριχθούν οι τοπικές κοινότητες, οι τοπικές αρχές ή γίνεται αυτό για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Και αυτό θα μπορούσαμε να το αναρωτηθούμε και για το Ταμείο Κοινωνικής Ένταξης. Πολύ συχνά τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται για πράγματα όπως οι επιστροφές και πολύ λίγο για την πραγματική κοινωνική ένταξη. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες ενδείξεις ή στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτού του καινούριου ταμείου προς το παρόν. Θα μείνω σε αυτά λέγοντας ότι συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια των συναδέλφων σχετικά με τις νομικές και ανθρωπιστικές υποχρεώσεις μας εδώ, αλλά και την ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Άτζα δεν είναι εδώ, ούτε η κυρία Μπιζότο, άρα ο Ντομινίκ Μαχτά θα μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία λεπτά και δύο ερωτήσεις. Ήδη συζητήσαμε, συζητούμε το θέμα αυτό και παρά την εξαιρετική δουλειά και την παρουσίαση των σημειωμάτων που έγινε, ε, θα πρέπει να πω ότι οι ε, κυρίες δεν κάλυψαν τις ανησυχίες μου. Καταρχά, μιλούμε για τι αριθμό. Ένα, ενάμιση εκατομμύριο, έξι εκατομμύρια, πόσοι. Το κόστος της επιχείρησης. 0,4, 0,6, 1% του ΕΠ. Ένα, 2, δέκα δις χωρίς να ξεχνούμε τα 3 με 6 δις το έτος που θα πρέπει να πληρώνουμε κατά 4 χρόνια στην Τουρκία. Μιλούμε για το ESF, μιλούμε για ειδικά κονδύλια, μιλούμε για νέα ταμεία σε σταθερό ποσοστό του προϋπολογισμού, αλλά έναντι ποιου. Εις βάρος τι πράγματος, της υποστήριξης των ανέργων μας, των νέων μας δεν έχω καταλάβει τις εξωτερικές σας παρατηρήσεις από τι αφαιρούμε. Και δύο θέματα τα οποία δεν αφαιρθήκατε μου φάνηκε. Πρώτον, πώς, θα, πώς εσείς διαφοροποιείτε ήδη μεταξύ των λεγόμενων πολιτικών προσφύγων και των οικονομικών προσφύγων γιατί μιλάτε για πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά μιλάτε για πολύ μεγαλύτερου αριθμούς από αυτού που θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και πολύ δυστυχισμένοι άνθρωποι που έχουν αφήσει πολλά πίσω τους. Μέλη τη οικογένεια τους, για παράδειγμα. Πώς φαντάζεστε δηλαδή ότι θα έχουμε κάποιε διατάξει για την ε, υποστήριξη των επιστροφών. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλέ. Από τι ερωτήσει που σας απευθύνθηκαν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Θα, κατα... θα κατανοήσουμε αν ε, επιλέξετε να μην δώσετε απαντήσει. Αν θέλετε απαντάτε. Ναι, όσο δυνατόν πιο σύντομα, παρακαλώ. Πολλά ενδιαφέροντα ακούστηκαν. Θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά καταρχάς με τη χρηματοδότηση. Από τα όσα γνωρίζω εγώ από τη δική μου ανάλυση, έχουμε τα εξή. Θα είναι μάλλον δύσκολο και χρονοβόρο να ειδηθεί ένα χωριστό χρηματοδοτικό μέσο το να ενταχθεί ένας τίτλος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πιστεύω ότι και έχοντας ακούσει βέβαια και ε, μέλη της ομάδας εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχει κίνδυνος και δέχομαι το επιχείρημα η χρηματοδότηση να χαθεί χρηματοδότηση θα μπορούσε να πάει σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα. Πάντως, προ το παρόν δεν υπάρχει συζήτηση συγκεκριμένη γι' αυτό, δεν έχει ενταχθεί τίποτα στην ανάλυση μα. Κόστος και σε ποιον θα προσφέρεται η εκμάθηση των γλωσσών και η κατάρτιση. Αυτά όλα έχουν ε, νομίζω κρυθεί από, την, ε, από τις στατιστικές τουλάχιστον, αλλά είναι και η απόφαση των πολιτικών πρόκειται για την επικουρική προστασία του διεθνούς δικαίου. Ο πρόσφυγας που προέρχεται από μια χώρα όπου δεν του επιτρέπουν οι συνθήκες να ζει με ασφαλή για την ζωή του, δεν μπορεί να αναγκαστεί να επιστρέψει στην χώρα αυτή. Εάν λοιπόν ένα 5% αναγνωρίζεται ως ε, πρόσφυγες καθαρά. Δεν ξέρουμε πώς είναι αυτοί που θα μείνουν για μεγάλο το χρονικό διάστημα επειδή θα παραμένουν οι κίνδυνοι που τους οδηγούν μακριά από τη χώρα τους. Και αυτό θα σήμαινε ευλογές επενδύσεις. Έστω και αν η άδεια παραμονής αρχικά προβλέπεται για ένα χρόνο και μετά γίνεται επανεξέταση των δικαιωμάτων. Γιατί μπορώ να πω ότι δεν έχω όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μου και για να απαντήσω και σε άλλε ερωτήσει. Εμείς εστιαστήκαμε κυρίω στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασία όχι στις, ε, στους επαναπατρισμούς. Και εκεί πέρα θα μείνουμε, ίσως μπορέσουμε να αναλύσουμε περαιτέρω κάποια άλλα ζητήματα. Ποια παραδείγματι είναι η διάρκεια κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ε, χώρες της Μεσογείου, που βρέχονται από τη Μεσόγειο από προβλήματα και ως προς τις δαπάνες και ως προς την λειτουργία και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας μπορεί να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πάντως χρειάζεται περισσότερο μελέτη και έρευνα η κατάσταση στις χώρες αυτές. Αυτά είναι τα κύρια σημεία νομίζω. Και ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε πάντα με την επιφύλαξη ότι είμαστε μόνο Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση και θα δώσουμε απαντήσει μόνο για θέματα του δικού μας πεδίου δράσεω. Για τον κύριο Μπενιφέη και, τις, ε, και το συνδυασμό χρηματοδότησης. Ευπρόσδεκτο το σχόλιο και απαντούμε ότι συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εντοπίσουμε στη λεπτομέρεια τις ανάγκες τους αλλά και τρόπους για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας. Γιατί όντως μπορούν να αξιοποιηθούν αρκετά διαφορετικά κονδύλια. Το ΦΕΟΓΑ, το ΕΜΙΦ, το ΦΕΑΔ, το κοινωνικό, τα μέρη του παγκοσμιοποίηση κτλ. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη για να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η χρηματοδότηση. Πρόκειται για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πολλές όμως ε, ε, πολλές δαπάνες καλύπτονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη και εμείς τα υποστηρίζουμε από πλευράς μας απευθείας. Για το αν θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ή λύση για το θέμα των δεξιοτήτων. Μας απασχολεί αυτό και προετοιμάζουμε το νέο θεματολόγιο δεξιότητων όπως υπόθηκε και νωρίτερα όπου λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες και ε, τα προσόντα και αυτό όχι μόνο για πρόσφυγες ή για άτομα έρχονται από τη μετανάστευση αλλά και για τους ε, πολίτες που ενδιαφέρονται για την κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια προσέγγιση λοιπόν για όλη την Ένωση που θα έχει να κάνει και με την αξιολόγηση δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των προσφύγων και προσόντων, που θα επιτρέπει την έκδοση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ή διαβατηρίου ε, δεξιοτήτων για τους πρόσφυγες. Αυτό λοιπόν το διαβατήριο δεξιοτήτων, όπως το έχουμε σχεδιάσει, μπορεί να μπει στο πλαίσιο του Europass, είναι μια λύση που εξετάζουμε. Μέσα από αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση που ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος έχει λάβει στη χώρα προελεύσεως. Μπορεί να γίνει κάποια επαλήθευση δεξιοτήτων, διευκρίνηση λεπτομεριών ε, μέσα από το σύστημα το εκπαιδευτικό ή με την επαγγελματική εμπειρία και βέβαια ιδιαίτερα όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες. Και εκεί θα κοιτάξουμε ποιες είναι οι ανάγκες, οι μαθησιακές και πάλι με έμφαση στη γλώσσα. Και αντίστοιχα θα έχουμε και ενημέρωση ε, πληρέστερη για τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες προελεύσεως. Αυτό σημαίνει στενή συνεργασία, εντατική συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων, επιπέδων αγοράς εργασίας, ε, αρχών αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων και άλλων. Μέσα στο νέο αυτό θεματολόγιο λοιπόν θα κοιτάξουμε και αυτά τα ζητήματα και αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τον πρόσφυγα αλλά και κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στην ανταλλαγή των πολλά υποσχόμενων νέων πρακτικών, όπω τι ονομάζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπα με προκλήσει στα κράτη-μέλη και προσπαθούν όσο το δυνατόν να απαντήσουν σε καταστάσει πρωτόγνωρε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε καλύτερες πρακτικές, με βέλτιστες πρακτικές, αλλά με πολλά υποσχόμενες πρακτικές. Αποκομίζουμε και από την εμπειρία των κρατών της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και από τις ε, νότιες χώρες. Εκδήλωση, σας είπα και νωρίτερα, προβλέπετε στην Ισπανία. Πάνω απ' όλα με αυτή τη διάσταση. Και εν τέλει, θα ήθελα να αναφέρω το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, έχει πολύ μεγάλη σημασία και κάποιοι από του ευρωβουλευτέ το έδειξαν. Έχουν εντό οι κοινωνικοί εταίροι ρόλο να διαδραματίσουν. Τον ρόλο αυτόν παίρνουν πολύ στα σοβαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερω ω προ τι δεξιότητε. Και έτσι επαναρχόμαστε στι δεξιότητε, γιατί μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να προσφέρουν κατάρτιση, είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα κάθε φορά, στην πράξη και μπορούν να εντοπίσουν ποιες είναι οι δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας. Άλλα ζητήματα που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσεως της ε, Γενικής Διευθυνσίας για την απασχόληση θα σχολιάσω. Ωστόσο σημειώνω πως υπάρχουν άλλες υπηρεσίες επιτροπής όπως η Γενική Διευθυνσία για τα Ιστορικά, η HOME, με πολλές δράσεις και κονδύλια. Σας ευχαριστώ. Θα κλείσει ο εισηγητής. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω την Επιτροπή για, όχι μόνο για αυτή την χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, αλλά για την συνεργασία που είχαμε ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες στην δουλειά την οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Από την συζήτηση βλέπουμε ξεκάθαρα κάποια θέματα που τίθενται στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων και κάποια θέματα που τίθενται από τους φιλοξενούμενους μας σήμερα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε λοιπόν τέτοιες απόψεις έτσι ώστε σαν κοινοβούλιο να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια τελική έκθεση χρήσιμη που θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες των εμπλεκομένων. Είναι σαφές και από τη συζήτηση που προηγήθηκε ότι για να ασχοληθεί κανείς με το θέμα αυτό απαιτείται καλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη εμπλοκή σε όλα τα θεσμικά επίπεδα ανάλογα με τις ευθύνες και επίσης εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είπα λοιπόν και στην βασική μου εισαγωγή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε για αρκετό καιρό ακόμα θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την ανταλλαγή των απόψεων και μετά την τελική υιοθέτηση ελπίζω της έκθεσής μας και θα συνεχίσουμε όλοι από κοινού όλα τα ευρωπαϊκά όργανα να συζητάμε σε θεσμικό επίπεδο αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο επανήλθε πολλές φορές και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν θέλουμε να είμαστε πράγματι πιο αποτελεσματικοί και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο τους υπάρχοντες πόρους και να βρούμε μεσοπρόθεσμα και κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια. Thank you. Ε, Σας ευχαριστώ. Η εξέταση των τροπολογιών είναι για τις 26 Απριλίου και η έγκριση 24 Μαΐου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Φτάσαμε λοιπόν στο... Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε στο ενδιάμεσο της μεγάλης απουσίας. Καλό βράδυ σε όλους.